Ladies Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι στη συνεδρίαση της ΑΦΚΟ. Με καθυστέρηση 15 λεπτών. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα θα συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης με βάση διάφορα έγγραφα εργασίας. Γνωρίζετε τις ε, συστάσεις των συντονιστών της 20ης Ιουνίου και της 13ης Ιουλίου, οι οποίες έχουν ε, ε, συμπεριληφθεί σε μια σειρά εγγράφων εργασίας. Συμφωνήσαμε όσον αφορά την μέθοδο εργασίας και το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση των εγγράφων. Ήδη νομίζω έχουμε παρουσιάσει τέσσερα τέτοια έγγραφα. Έξι μάλλον, και δύο απομένουν. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο. Το ένα έχει να κάνει με την εμβάθυνση της ΟΝΕ, της Mercedes Πρέσο και ΕΜΟΥ. Και το δεύτερο έγγραφο εργασίας έχει να κάνει με την δομή και, την, και τον τρόπο εργασίας του Συμβουλίου του κυρίου Γιαστόφσκη και της κυρίας Ταπανέλ. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι διαθέσιμο στο σύνολό του. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε αυτά που συμπεριλαμβάνει αυτή τη στιγμή το έγγραφο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο έγγραφο εργασίας. Δίνω πέντε λεπτά στον κάθε ομιλητή και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το έγγραφο προβληματισμού για την εμβάθυνση της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εμού και της Μερσέντες. Μερσέντες, αν δεν έχει αντίρρηση, θα σου δώσω πρώτα το λόγο και μετά θα μιλήσω εγώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, αυτά τα έγγραφα εργασίας ε, είναι καρπός ε, σύνθετης δουλειάς, διότι όπως γνωρίζετε περιλαμβάνει ένα τμήμα το οποίο συνοψίζει τις ε, θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό στο παρελθόν, κυρίως για τις ε, πτυχές ε, θεσμικού χαρακτήρα που έχουν βέβαια άμεση σχέση και με τα υπόλοιπα. Το πρώτο τμήμα, κατά πάσα πιθανότητα, χρειάζεται και κάποιες ε, προσθήκες, διότι προσφάτως αντιλήφθηκα ότι ουσιαστικά λάβαμε υπόψη τις εκθέσεις που έγιναν στην Επιτροπή μας, ενώ όπως είναι γνωστό Υπάρχουν και κάποιες εξίσου σημαντικές εκθέσεις οι οποίες ε, ε, είναι και αυτές σημαντικές από θεσμική σκοπιά από άλλες επιτροπές, κυρίως από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, την τρίτη έκθεση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αντιλήφθηκα ότι δεν ε, αναφέρεται παρκώς ε, σε σχέση και με τη σημασία των θεμάτων ε, των οποίων άπτεται ακόμα και θεσμικού χαρακτήρα. Αυτό βέβαια όμως μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να βελτιώσουμε το σκέλος που αφορά το πρόσφατο παρελθόν διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για εκθέσεις πάρα πολύ πρόσφατες. Το τμήμα το οποίο ε, καταρτήσαμε με τον συνάδελφο Πάιπερ αφορά το ε, εγγύης αλλά και το μακροπρόθεσμο μέλλον για το θέμα αυτό. Όπως ε, γνωρίζετε βρισκόμαστε σε μια ε, στιγμή γεμάτη προτάσεις διότι η Επιτροπή μέσω της Λευκής Βίβλου, μέσω και ενός πολύ συγκεκριμένου εγγράφου στο οποίο γίνεται μια ε, εις βάθος ανάλυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και μέσω και των προτάσεων που έχουν ανακοινωθεί και οι οποίες ε, λογικά θα πρέπει να εγκριθούν και από εκεί και πέρα να μας γνωστοποιηθούν ε, το Δεκέμβριο έγινε μια διεξοδικότατη εμβριθής ε, δουλειά και επομένως οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτό το υπενθυμίζουμε και στο έγγραφο και τις αρμοδιότητες ε, των ε, πιο εξειδικευμένων επιτροπών πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής ΕΚΟΝ, αλλά και κάποια θεσμικά θέματα στα οποία προσπαθούμε να εμβαθύνουμε τη δουλειά μας. Δεν θα τα πω όλα γιατί θέλω να αφήσω και κάτι να παρουσιάσει ο συνάδελφος, αλλά εγώ νομίζω ότι θα ήθελα να σταθώ στις αρχές που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές ε, για να εμβαθύνουμε στα θέματα τα οποία αφορούν ε, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη δημοκρατία, την ευθύνη και την αλληλεγγύη. και πιο συγκεκριμένα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο οποίος πρέπει να είναι εγγυημένος για τις ε, ε προόδους που θέλουμε να επιτύχουμε και προσπαθούμε να επεξεργαστούμε. Εδώ λαμβάνουμε υπόψη μας και τις προτάσεις του Προέδρου Γιούνκερ, τα όσα ανακοίνωσε και αυτά θα περιλαμβάνουν δύο πτυχές. Η μία πτυχή θα αφορά μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να γίνει τροποποίηση των συνθήκων ε, που από πλευρά μας θα πρέπει ε, να αποτελούν και προτεραιότητα και για λόγους ε, χρονοδιαγράμματος αλλά και για να υποβληθούν τα διάφορα έγγραφα τα οποία ε, μας υπέδειξαν, δηλαδή τι μπορεί να γίνει χωρίς τροποποίηση των συνθήκων και ε, στη συνέχεια πιθανώς ε, και τροποποίηση των συνθήκων, αλλά και εντό των συνθήκων που έχουμε ενισχύει αυτή τη στιγμή, που νομίζω ότι όπω αποδείξαμε με το έγγραφο που κάναμε με τον συνάδελφο Μπροκ, υπάρχει περιθώριο για να αυξηθεί η δημοκρατική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, στις επόμενες προοπτικές έχω την εντύπωση ότι μία πρόταση για ένα κονδύλι στον προπολογισμό, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή η οποία θα είναι ε, αφιερωμένη στην ε, Ευρωζώνη. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να είναι μια γραμμή η οποία θα στοχεύει σε επενδύσεις προφανώς, αλλά επίσης όπως ανακοινώθηκε και θα μπορεί να βοηθήσει και τις χώρες οι οποίες ε, προετοιμάζονται να ενταχθούν στο ευρώ, ιδίω εκείνε οι οποίε είναι διατεθειμένε να ακολουθήσουν ένα πολύ συγκεκριμένο χάρτη πορεία ε, για ε, την ένταξη στην ευρωζώνη και στο ευρώ. Εκφράζουμε και το γεγονός ότι είμαστε ευνοϊκά διακείμενοι ε, στην ιδέα ενός ε, Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών Θεμάτων, όπως προτάθηκε και στο έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πιο συγκεκριμένα, από θεσμική σκοπιάς, εάν αν ο πρόεδρος της Ευρωζώνης είναι κάποιο ο οποίο ταυτόχρονα θα είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, θεωρούμε ότι θα βελτιωθεί ουσιαστικά και η δυνατότητα ελέγχου από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, Ε, θα έχει επιπλέον αρμοδιότητες διότι ο πρόεδρος και το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα είναι υπόλογος έναντι του Κοινοβουλίου. Βεβαίως ε, όσον αφορά το ρόλο αυτό του Υπουργού θα συζητηθούν και οι προτάσεις που θα προκύψουν. Όσον αφορά τους ίδιους πόρους για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την εντύπωση ότι αυτή είναι θεμελιώδης ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη για ένα πιο ανεξάρτητο προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούμε ότι αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη της βελτίωσης της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης και αντιστοίχως ε, και ε, της λογοδοσίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πρέπει να βελτιωθεί και για αυτό το συγκεκριμένο. Ε, αναφέρουμε το θέμα της εξωτερικής εκπροσώπησης της Ευρωζώνης. Ε, αναφερόμαστε επίσης και στο ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί και από πλευράς ελέγχου, από πλευράς των Εθνικών Κοινοβουλίων. τα οποία θα πρέπει να βελτιώσουν και την εθνική διάσταση της συζήτησης και της αξιολόγησης και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να βελτιωθεί ε, όχι απαραίτητα με αλλαγή των συνθήκων, αλλά ε, μέσω μιας πιθανής διοργανικής συμφωνίας. Νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ και να αφήσω στο συνάδελφο να σας αναπτύξει τα υπόλοιπα θέματα και φυσικά ε, και για παρατηρήσεις ε, για το έγγραφο, αλλά σίγουρα ένα τμήμα του εγγράφου δεν ε, θα το παρουσιάσω για να μπορέσουμε να μοιραστούμε και αυτά τα καθήκοντα, όχι μόνο όσον αφορά τη γενικότερη παρουσίαση, αλλά και για τα διάφορα σημεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Τότε πρόεδρος θα μου δώσω και εμένα το λόγο. για να σχολιάσω το έγγραφο προβληματισμού. Η Μερσέντες τα είπε όλα, λίγο πολύ. Ε, μπορώ όλες να επιβεβαιώσω τα περισσότερα από όσα είπε. Δύο σημεία του εγγράφου δεν ανέφερε και θα τα σχολιάσω εγώ. Από τη μία περιμένουμε καλύτερη σύνδεση αυτών που κάνουμε εδώ στην ΑΦΚΟ, στο Κοινοβούλιο, στις πολιτικές ομάδες, με αυτά που γίνονται στην ΕΚΟΝ, διότι οι εκθέσεις της ΑΦΚΟ δυστυχώς ε, ψηφίστηκαν με πολύ ασθενή πλειοψηφία. και η έκθεση Φερχόφστατ πήρε 280 ψήφους από τους 750 βουλευτές. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να θεωρηθεί ε, μια στιβαρή βάση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τη στιγμή που υπάρχουν ε, τέτοιες διαφωνίες. Άλλο θέμα το οποίο είναι θεμελιώδου σημασίας σε σχέση με τον προϋπολογισμό τα δημοσιονομικά, την θετική οικονομική εξέλιξη. Είναι αυτό που τονίζουμε στην έκθεση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει όλη την ευθύνη. Η βάση για την πολιτική, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για δημοσιονομικά και χρέος, ε, βρίσκεται στα κράτη-μέλη. Άλλο ένα θέμα στο οποίο επίσης συμφωνούμε και που δεν θα αφήσουμε να μας διχάσει είναι η πρόταση για προϋπολογισμό της Ευρωζώνης και συνέλευση της Ευρωζώνης. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει προϋπολογισμός ο οποίος να διατίθεται στα κράτη της Ευρωζώνης ε, και στα άλλα κράτη, τα opt-in κράτη. Τέταρτη παρατήρηση. Το θέμα της αύξησης των ιδίων πόρων, ε, διότι ε, δεν είναι σωστό κάθε δύο χρόνια να πρέπει να κάνουμε παζάρια για να πετύχουμε αύξηση των πόρων μας, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Όσον αφορά τον Υπουργό Οικονομικών, ε, αγαπητή κυρία Μπρέσο, δεν ξέρω πόσες φορές το συζητήσαμε αυτό. Χρειαζόμαστε περιγραφή των καθηκόντων ενός τέτοιου Υπουργού οικονομικών της Ευρωζώνης. Επικροτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει τη δημιουργία της θέσης αυτής. Πιστεύουμε σίγουρα ότι ε, τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Δεν ε, απαιτούμε όμως Υπουργό Οικονομικών ε, της Ευρωζώνης στο έγγραφο. Αυτό παραμένει ανοιχτό και θα πρέπει να το συζητήσουμε. δεν αναφέρεται στο έγγραφο όπως είπα. Το αφαίρεσαμε από το κείμενο και ε, κυρία Περές ε, θα μπορέσετε να το σχολιάσετε αυτό μετά. Συζητήσαμε μήπως θα είναι πιο χρήσιμο να διατηρήσουμε ως επικεφαλής της Ευρωζώνης έναν Υπουργό Οικονομικών κράτους μέλους, διότι έτσι η σχέση με τα κράτη-μέλη, η επαφή με τα κράτη-μέλη θα είναι ισχυρότερη. Μπορεί όμως να υπάρχει και μια ενδιάμεση λύση, την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να έχουμε το Κοινοβούλιο μαζί μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε μια ψηφοφορία με αποτέλεσμα 50-50% διότι τότε τα κράτη-μέλη θα μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό προσπαθήστε να πετύχετε και την ε, συμμετοχή των συναδέρφων σας ε, όλων στις ψηφοφορίες στην ΑΦΚΟ. Επίσης, όσον αφορά τον ε, κώδικα σύγκλησης, η κυρία Πρέσο αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να οργανώσουμε ακρόαση για να εμβαθύνουμε στο μέλλον της ΟΝΕ. Εάν προχωρήσουμε στην εμβάθυνση, φέρουμε ευθύνη για τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών δεν επιτρέπεται να προχωρήσουμε τόσο στην εμβάθυνση ώστε ε, μέρος των κρατών μελών να παραμείνει απ' έξω, πιθανότατα για πάντα. Τα επόμενα βήματα εμβάθυνσης θα πρέπει να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Να μην κλείσουμε την πόρτα. Γι' αυτό καλύτερα να προχωρήσουμε αργά με μικρά βήματα και να πετύχουμε τη συμμετοχή όλων, αντί να βιαστούμε και να διχάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωεκλογές επίκυνται και η ΑΦΚΟ φέρει μεγάλη ευθύνη να κοιτάξει και την Βόρεια Ευρώπη και την Νότια και την Ανατολική και τη Δυτική και να επιδιώξει λύσεις που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όχι λίγων αλλά όλων. Αυτές οι δύο τελευταίες ήταν δικές μου προσωπικές παρατηρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο προβληματισμού. Όλα τα υπόλοιπα όμως συμπεριλαμβάνονται και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την συνάδελφο την κυρία Μπρέσο διότι καταφέραμε να βρούμε κοινή βάση. Είχαμε μακρές συζητήσεις, αλλά καταφέραμε να βρούμε κοινή βάση πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να, να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Κλείνω τη δική μου παρέμβαση. να ακούσουμε τους συναδέλφους ή να προχωρήσουμε στο άλλο έγγραφο. Να προχωρήσουμε στο επόμενο έγγραφο. δομή και μέθοδο εργασία ε, του Συμβουλίου. Ο κύριο Ουγιαστόφσκι έχει πρώτο το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το έγγραφο το οποίο αναφέρεται στην μέθοδο εργασίας του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μία πρόταση την οποία έχω καταθέσει εγώ προσωπικά. Αυτό το οποίο περιμένω είναι η συμβολή του κυρίου Τσαπαρντέλ. Ελπίζω πως τελικά θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι η δική μας κοινή προσπάθεια και με μεγάλη χαρά περιμένω προτάσεις και ιδέες από πλευράς του. Πρέπει να σας πω πως εκτιμώ ιδιαίτερα τα όσα μόλις ακούσαμε από τον προηγούμενο μιλητή, γιατί πιστεύω κι εγώ πως καλύτερη προσέγγιση είναι μια συνετή προσέγγιση της όλης διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το δικό μου έγγραφο βασίζεται στην εξής σκέψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή θεσμική επανάσταση. Χρειάζεται απλώς μία ανοικοδόμηση της αμοιβαία εμπιστοσύνης σε πολλά επίπεδα και αυτό συμπεριλαμβάνει και την ανάκτηση της εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δηλαδή, σεβασμός για την αυτονομία και ξεχωριστή φύση κάθε διαφορετικού θεσμού. Η αλήθεια είναι πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τα δικά του δικαιώματα, το δικό του ρόλο και ε, φανταζόμαστε πως τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα θα δεχθούν τα παραπάνω. Προφανέστατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν κάτι αντίστοιχο από εμάς. Θα πρέπει δηλαδή να σεβαστούμε και εμείς την αυτονομία του Συμβουλίου, όπως επίσης και το γεγονός πως έχει κάποιο είδους εσωτερική ευελιξία που εφαρμόζει. Το Συμβούλιο λειτουργεί ε, σε πολλαπλούς ε, σχηματισμούς και ενδεχομένως κάποιοι ακόμα δεν έχουν καν εμφανιστεί. Αυτό είναι πολύ θετικό για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο καθηγητής κ. Χάινολτ κατέθεσε πρόταση και αυτό μέσω μιας μελέτης για ένα νέο σχηματισμό ε, που θα συμπεριλάβει την αστική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Το Συμβούλιο όμως χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του να έχει αυτό το βαθμό της ε, εσωτερικής ευελιξίας. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο την εξής πρακτική. Γιατί σε επίπεδο θεσμικών εργάνων υπάρχει και η εξής μέθοδος εργασίας. οι προτάσεις των κρατών μελών. Γιατί ας πούμε έχουμε την πρόταση, έχουμε το non-paper της Σουηδίας για την εξωτερική πολιτική. Νομίζω πως στο έγγραφο αυτό προτάθηκε μια νέα μεθοδολογία εργασίας για το Συμβούλιο ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκεί στηρίχτηκε η Σουηδία από τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, τις κάτω χώρες και το Βέλγιο. Και η πρόταση ήταν η εξής να βρεθούν κάποιες νέες ε, εύκολες και πρακτικές στην εφαρμογή τους λύσεις χωρίς να αλλάξουν οι κανόνες ψηφοφορίας στο Συμβούλιο και πιο συγκεκριμένα να υπάρχει η δυνατότητα περισσότερο μεγαλύτερη μεγαλύτερης και πιο εντατική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ ΙΠΕΞ και με... μαζί με την ανώτατη εκπρόσωπο την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό στα πλαίσια των όσων κάνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Κάτι ακόμα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ε, να δούμε πώς θα λειτουργήσει καλύτερα ε, το τρίο προεδριών. Έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, πιο ολοκληρωμένη συνεργασία πριν ξεκινήσει κάποιο κράτος στην προεδρία του και αυτό έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συνέχεια από τη μία προεδρία στην επόμενη. Κάτι που ακόμα που προτείνω είναι να διευρύνουμε την διαφάνεια τη διαφάνεια σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αποδείξει πως δεσμεύεται υπέρ της διαφάνειας και να ε, επιτελεί το έργο του με υποδειγματικό ε, τρόπο. Αυτά με χαρά περιμένω τη συζήτηση που θα κάνουμε μεταξύ μας και συμπερασματικά θα δηλώσω το εξή. Πρέπει να ανακτήσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Χρειάζεται βέβαια να ανακτήσουν ε, ε, την εμπιστοσύνη τους ή τα θεσμικά όργανα με απόλυτο σεβασμό των ιδιαζόντων τους χαρακτηριστικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Ταπαρδέλ θα ήθελα να συμπληρώσει. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου, κυρία Ταπαρδέλ. Now it's functioning. Okay, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω και τον συνεισηγητή και με μεγάλη χαρά διαπιστώνω πως σήμερα έφτασε η ώρα να συζητήσουμε αυτό το έγγραφο ε, το οποίο έχει να κάνει με πολύ σημαντικά ζητήματα που άπτονται της μεθοδολογίας εργασίας του Συμβουλίου. Βεβαίως ακόμα είναι η υποσυζήτηση η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης και το έγγραφο προβληματισμού δεν ε, αναφέρεται συγκεκριμένα στο θέμα αυτό. Δηλαδή δεν μιλάς για κάποια θέματα τα οποία και την Ευρωζώνη και την ΟΝΕ τη αφορούν ιδιαίτερα. Χρειαζόμαστε καλύτερη διακυβέρνηση, αλλά αυτό πρέπει να συμβεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλουμε και μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση. Να σας πω τώρα για τα θέματα του Συμβουλίου πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμα δεν έχει ετοιμάσει καμία έκθεση που να αναφέρεται συγκεκριμένα στη μεθοδολογία εργασία του Συμβουλίου. Όμως, κάποτε παρουσιάσαμε μια εποχή σε ε, μία σειρά από συστάσεις ε, με προτάσεις για τροποποιήσεις και για αναδιάρθρωση και αυτό στα πλαίσια της αναθεώρησης της συνθήκης της Λισαβόνας. Άρα λοιπόν αυτό που θα κάνω τώρα είναι να παρουσιάσω μία σειρά από σχόλια και σκέψεις που έχω σχετικά και αργότερα θα παρουσιάσουμε και την ε, τελική μορφή του εγγράφου μαζί με τον συνεισηγητή μου. Η συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιγράφεται από τις διατάξεις που έχουμε στη συνθήκη και πάντα με απόλυτο σεβασμό των αμοιβαίων αρμοδιοτήτων, της θεσμικής ισορροπίας, του θεμητού και της θεμητής συνεργασίας, της κοινοτικής μεθόδου, όπως επίσης και του σεβασμού των ευρωπαϊκών αρχών. Όταν ετέθη σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνα και με τις μεγαλύτερες αρμοδιότητε που εκεί εκχωρήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συνεργασία διαστρώθηκε, δομήθηκε με πιο συγκεκριμένο τρόπο και απέκτησε μεγαλύτερη ένταση. Και αυτό λόγω ε, των νομοθετικών ε, δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ελέγχου που απέκτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πάντα λόγω της αύξησης των διαδικασιών ε, συναπόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τη συνθήκη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, ε, είναι ίσοι και οι συμφωνίες γίνονται χωρίς να υπάρχει η πολιτική υποχρέωση αλλά βασιζόμενη στην αυτονομία των θεσμικών οργάνων και στο σεβασμό αλλήλων. Και η το Better Legislation, για παράδειγμα, είναι μια σχετική, ε, ένα σχετικό παράγραμμα, όπως επίσης προγραμματισμός και το θεματολόγιο ε, των όσων συζητιούνται κάθε χρόνο. Έτσι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το ετήσιο δράσης, στο οποίο για το οποίο συνεργαζόμαστε όλοι, με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη συνοχή. Εδώ λοιπόν αυτό που είναι σημαντικό είναι ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτός που γίνεται επίσημα και αυτός που γίνεται ανεπίσημα για τις προτεραιότητες του προγράμματος, για να είναι πιο αποτελεσματικό το θεματολόγιο και για να απλουστευτεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων. Γιατί εγώ είμαι πεπισμένη πως μόνο με μέσω του διαλόγου και τη συνεργασίας θα γίνουμε πιο ορατοί και θα έχουν ε, τη δυνατότητα να μας γνωρίσουν καλύτερα οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και έτσι θα πετύχουμε και εμείς τους στόχους μας και θα εξασφαλίσουμε πως υπάρχει συνεχή, πως υπάρχει συνέχεια σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Σχετικά τώρα για τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νομίζω πως κάτι τέτοιο, ναι, θα βελτίωνε τις ε, επιδόσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η ιδέα αυτή, ξέρετε πως δεν έχει πρικοδοτηθεί με αρκετά επιχειρήματα. Είμαστε σε μια πρώτη φάση ακόμα και για τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των καρτών μελών και εκεί ακόμα υπάρχουν κάποια κενά. Για τη λήψη αποφάσεων, αν δούμε εδώ τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι, απο... αποφάσει στο Συμβούλιο, θα διαπιστώσουμε πω η συνθήκη τη Λισαβόνα ορίζει ποιοι είναι οι χώροι κατά του οποίου μπορούν να αποφασίσουν με ειδική πλειοψηφία ή με ομοφωνία. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγή ε, του τρόπου λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε από την ομοφωνία να περάσει κανεί στην ειδική πλειοψηφία κτλ. Δηλαδή, ε, μέσω ας πούμε της συγκεκριμένης ρήτρα θα μπορούν κάποια κράτη-μέλη μετά από ε, σχετική, σχετικά αιτήματα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να αλλάξουν αυτή την ψηφοφορία και να μην γίνεται πλέον με ομοφωνία αν κριθεί αυτό απαραίτητο. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει εδώ να εξετάσουν κατά πόσο είναι σωστό στις περιπτώσεις αυτές και σε διαφορετικούς κλάδους να έχουμε αποφάσει με ειδική πλειοψηφία γιατί βεβαίως χρειαζόμαστε συνενετικές αποφάσεις, έτσι ώστε να μην προχωρήσουμε σε ένα κατακαιρματισμό σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντικό να σταθούμε πολύ συνετά στο, θέμα αυτό της ενισχυμένης συνεργασίας. Πρέπει να σας πω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να ακολουθήσει ε, όσο το δυνατόν πιο αλληλέγγυα και ενιαία στάση στο θέμα της λήψης αποφάσεων και μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο να φεύγει από τον κανόνα αυτό. Για την δομή του Συμβουλίου συμφωνώ με τον εισηγητή. Ο βασικός του νόμος που διέπει ε, αυτή τη λειτουργία του Συμβουλίου είναι ε, αυτός για την αυτονομία των εσωτερικών διευθυντήσεων. Αλλά, ξέρετε, πως είναι πολύ βασικό να αποφεύγουμε επικαλύψεις παραλληλισμούς και ε, δυσλειτουργίες. Για το τρίο των Προεδριών και για το θέμα που έχουν στο Συμβούλιο νομίζουμε πως θα πρέπει αυτό να ενισχυθεί και να έχουμε κάτι αντίστοιχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, για μεγαλύτερη συνοχή, να σας πω πως θα πρέπει το θεματολόγιο και ο προγραμματισμός να έχουν περισσότερη διαφάνεια και να είναι αποτέλεσμα συνένεσης και οι προτεραιότητες. Και χρειαζόμαστε και ε, πολιετή προγραμματισμό, κάτι το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει, κάτι το οποίο κρίνω ήδη πολύ θετικά, γιατί με τον τρόπο αυτό ε, καταφέρνουμε να παγιώσουμε καλύτερα ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για το πώς ε, το τρίο εδριών μπορούν να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σας πω πως μόνο στη Ρουμανία, για παράδειγμα, που προετοιμάζεται για την Προεδρία της το 2019, το πρώτο εξάμεινο, ήδη συζητάμε το θέμα αυτό και έχουμε λάβει υπόψη πάρα πολλές από αυτές τις παρατηρήσεις. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν που θα εξυπηρετεί και θα υπηρετεί τους πολίτες πιο ανοιχτή, πιο διάφανη και που θα σέβεται περισσότερο τις ε, βασικές αρχές θα συνεισφέρει στο να ανακτήσουμε την ε, εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τη στηρίξει περισσότερο το ευρωπαϊκό κοινό. Η υποχρέωση διαφάνειας είναι κάτι το πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της διοικητικής και πολιτικής διαδικασίας που ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνης, είναι πιο ανοιχτέ οι διαδικασίες στο Συμβούλιο και η διαφάνεια σαφώς έχει αυξηθεί. Έχει μεγαλύτερη πρόσβαση το κοινό στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Επίσης, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έφερε ένα θέμα αυτή τη στιγμή σε συζήτηση που είναι η καταχώρηση στο Μητρό διαφάνεια και μέσω αυτού του Μητρώου θα μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις μεταξύ υπηρεών και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, όπως επίσης διαφόρων φορέων και οργανώσεων που εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω στο Συμβούλιο ήδη ξεκίνησαν για να δημιουργήσουν μια πύλη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι κατεξουσιοδότηση πράξεις. Έτσι ώστε και εκεί να τακτοποιηθεί το θέμα. Επίσης, μία τέτοιου είδους πύλη για την κοινή νομοθεσία που θα κάνει κάτι αντίστοιχο. Παρ' όλα αυτά, τα μέτρα αυτά ε, ε, έχουν σκοπό μεν να αυξήσουν τη διαφάνεια, αλλά δεν είναι και τέλεια. Ε, θα το αφήσω εδώ και θα ακούσω και τους συναδέλφους και όπως είπα και στην αρχή ξεκινώντας θα συνεργαστούμε με τον συνεισηγητή έτσι ώστε τα έγγραφα τα οποία λείπουν να τα καταθέσουμε εμπρόθεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ταπαρντέλ, όντω ε, προσθέσατε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Και τώρα θα πρέπει να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές ε, και για τα δύο εγγραφά εργασίας. Ποιος θέλει το λόγο παρακαλώ. Η κυρία Μπερές είναι στον κατάλογο αλλά δεν είναι εδώ. Εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε εδώ με τα έγγραφα εργασία. Θα μιλήσω γερμανικά τώρα. Επόμενα βήματα. Πρώτον, τα έγγραφα προβληματισμού, το έγγραφο προβληματισμού για το Συμβούλιο θα συμπληρωθεί με τις παρατηρήσεις της κυρία Σταπαρδέλ. Β, Πολύ σύντομα θα υπάρξει σύνοψη των εγγράφων προβληματισμού. Όλα τα έγγραφα αυτά σχετίζονται με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, θα διαβαστούν στους συντονιστές με τις παρατηρήσεις που ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τέταρτον, θα αποφασιστεί τι είδους εκθέσεις θέλουμε με βάση τα έγγραφα προβληματισμού για να υποβάλουμε στην Ολομέλεια ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης. Θα κλείσουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή. Ε, κύριε Σεπφλίν, παρακαλώ, το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, περίληψη, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε ίσως ότι θα γίνει μια σύνοδο στις 23 Φεβρουαρίου που θα ασχοληθεί με πολλά από τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση και δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσαμε να καταρτήσουμε κάποιο έγγραφο ε, ελπίζοντας να μπορέσουμε να επηρεάσουμε και εμείς κάπως τη συζήτηση. Ε, δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνος, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε και τις ιδέες μας εκεί. Θα ήταν ο κατάλληλος χώρος. Δυστυχώς, δεν έχω την αρμοδιότητα να σας απαντήσω, θα ήταν κρίμα όμως κατά τη γνώμη μου εάν ως ΑΦΚΟ ή ως Ευρωκοινοβούλιο δεν ε, συμβάλλουμε στη συζήτηση πριν από αυτή τη διάσκεψη κορυφής. Είναι λοιπόν καλή πρόταση και πολύ ευχαρίστως ε, θα την ε, διαβιβάσουμε στους συντονιστές. Να έχουμε δηλαδή μία συνοπτική έκθεση ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε τις θέσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση αυτή. Ωραία, σύντομο διάλειμμα. Κυρία Μπρέσο, παρακαλώ. Ε, αν Αν και λυπάμαι διότι είναι δύσκολο να γίνει η συζήτηση σε απουσία της Πρόεδρου, διότι οι προτάσεις για τα έγγραφα αυτά ε, ήρθαν από την ίδια και τα είχαμε συζητήσει και στις συνεδρίες των συντονιστών. Από αυτά που κατάλαβα, τα έγγραφα δεν θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια, αλλά επίσης δεν θα ψηφιστούν και στην Επιτροπή. Πρόκειται για έγγραφα ε, μέσα των οποίων εμβαθύνουμε σε κάποια θέματα και ήδη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν εκφράσει την άποψή τους για τα θέματα αυτά και υπάρχουν και προτάσεις για να εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά θα διακόψω. E ένα δευτερόλεπτο και τελειώνω. Επ' αυτή της βάση, λοιπόν καταλήξαμε ότι σε επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών θα γίνουν κάποιες προτάσεις για να χρησιμοποιήσουμε ίσως ένα τμήμα αυτών των εργασιών για εκθέσεις οι οποίες μπορούσαν να είναι εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας, δεν έχουμε βέβαια και πολλές τέτοιες. Θα μπορούσαν να είναι εκθέσεις εφαρμογής για τα θέματα επί των οποίων έχουμε ήδη ψηφίσει. και ψηφίσματα ή αντίστοιχα πράγματα. Απλώς ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται να υπάρχει διαδικασία ψηφοφορίας, γιατί αλλιώς θα πρέπει να ξεκινήσει και διαδικασία κατάθεσης τροπολογιών και στη συνέχεια να ψηφίσουμε. Αλλά δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα έγγραφα ως βάση για να γίνουν προτάσεις ε, πρωτοβουλίας της Επιτροπής ε, οι οποίες ε, θα αποφασιστούν αλλά ακόμα δεν έχουμε διαπιστώσει ποιες είναι. Ήρθε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς τώρα, επομένως θα σιωπήσω, θα ξαναδούμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή στο μέλλον. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Ευχαριστώ που προσκαλέσατε και την Επιτροπή μου και την υποφαινούμενη για να μοιραστεί αυτό το απόγευμα μαζί σας, μαζί με τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερμανς. Και τώρα, επειδή λείπει και η πρόεδρος της Επιτροπής σας ε, για κάποιο λόγο, Ευχαριστώ λοιπόν που μας δίνετε την ευκαιρία να είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα για να συζητήσουμε τον κανονισμό ε, για την πρωτοβουλία των πολιτών που εξετάσαμε και εμείς από πλευράς Επιτροπής μας. Ε, προτείναμε και κάποιες βελτιώσεις ε, στη γνωμοδότηση προς την νομοθετική έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της ΑΦΚΟ που έγινε το Σεπτέμβριο φέτος. Με χαρά διαπιστώνω ότι πολλά από τα σημεία που θίξαμε εμείς στην Επιτροπή μας αναφέρονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και είμαστε ευγνώμονες. Είμαι πεπισμένη ότι μετά από τα όσα θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο νέος κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών θα ε, προσφέρει πολύ πιο πρακτικές και ένα ε, πτυχές και ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι πιο φιλικό προς το χρήστη για να υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τελείως διαφορετικό από την κατάσταση που ισχύει σήμερα. Με αυτό λοιπόν ως σημείο κίνησης ας ξεκινήσουμε τώρα δίνοντας το λόγο βεβαίως στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερμαντς. Φράνς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εδώ σήμερα, διότι πραγματικά χαίρομαι που σας παρουσιάζω την πρότασή μας για την αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού για την πρωτοβουλία των πολιτών. Ιδίως διότι ε, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό με αρκετούς από εσά ε, ιδιαίτερα έντονα τους τελευταίους ένα-δύο μήνες. Το άρθρο 11 της συνθήκης οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν απευθεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση. Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από ένα εκατομμύριο πολίτες και άνω, από σημαντικό αριθμό κρατών μελών και η διάταξη αυτή είναι μεταξύ των δημοκρατικών αρχών της Ένωσή μα και πιστεύω ότι είναι μία από τι πιο θετικέ εξελίξει της ε, ε, συνθήκης που οδήγησε στη συνταγματική συνθήκη. Αυτό που διακρίνει τη δημοκρατία ως πολιτικό σύστημα είναι η δέσμευση για πολυφωνία και ε, ο συνδυασμός πληθώρας μέσων και διαδικασιών είναι αυτός ο οποίος κάνει το σύστημα δημοκρατικό με την πλήρη έννοια του όρου. Το αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημοκρατικοί θεσμοί έχουν ουσιαστική ανάγκη να έρχονται συνεχώς σε επαφή με τους πολίτες και αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους. Αλλά η συνθήκη μας ξεχωρίζει την πρωτοβουλία των πολιτών ω ένα πολύ σημαντικό δίαπλο για να επιτευχθεί αυτό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για το δημοκρατικό βίο της Ένωσης ε, η πρωτοβουλία των πολιτών να γίνει ένα ζωντανό μέσο το οποίο θα λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Να ξέρουν οι πολίτε ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να προτείνουν τι ιδέες του και να εισακουστεί η φωνή του. Η ε, πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να είναι εύκολο και να μην είναι μια διαδικασία γεμάτη γραφοκρατικά προσκόμματα. Εδώ και πέντε χρόνια λειτουργεί το σύστημα. Η πρωτοβουλία των πολιτών είχε κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Πάνω από 8 εκατομμύρια πολίτες συνολικά έχουν υποστηρίξει τις 47 πρωτοβουλίες που κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέσσερις από αυτές τις πρωτοβουλίες πέρασαν το κατόφλι των 1 εκατομμύριων πολιτών και ξεκίνησαν τη διαδικασία ώστε να γίνουν ενωσιακοί πολιτική. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προτάσεις των πολιτών και προτείνουμε ε, να ε, προτείνουμε ε, πολύ σύντομα μία αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό σε συνέχεια της πρότασης πρωτοβουλίας των πολιτών. Ε, μέχρι τον Ιανουάριο θα απαντήσουμε επίσης και για την πρωτοβουλία για να σταματήσει το γλυφοσάτ, το οποίο η γλυφοσάτη δεν αποτελεί μόνο πρόταση για τη γλυφοσάτη, αλλά γενικότερα για τα φυτοφάρμακα. Ε, η πρωτοβουλία όμως των πολιτών ως μέσο για τη συμμετοχική δημοκρατία έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες τις οποίες δεν έχουν εκμεταλλευτεί οι πολίτες μέχρι τούδε. Δεν είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν την ύπαρξή τους, δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι υπογράφουν πρωτοβουλίες ε, και ακόμα και κάποιοι που πιθανόν ενδιαφέρονται ε, τους αποτρέπει ε, η, η γραφειοκρατία και αντιμετωπίζονται πολλά προσκόμματα και πρακτικές δυσκολίες όπως διαπιστώθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τον Νοέμβριο του 2014 η Επιτροπή μας έλαβε πολύ συγκεκριμένα βήματα βάσει του παρόντος πλαισίου και προσπαθεί να προχωρήσει ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Τώρα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά την καταχώρηση των πρωτοβουλειών πριν τη συλλογή των υπογραφών, λαμβάνονται αποφάσεις σε επίπεδο του Σώματος των Επιτρόπων και επιτρέπουμε και μερική καταγραφή των πρωτοβουλειών, κάτι που είναι σημαντική αλλαγή και γίνεται διάκριση ώστε μπορούμε να κατανοήσουμε ποιο τμήμα της πρωτοβουλίας είναι παραδεκτό και ποιο όχι να σας αναφέρω και τα πιο σημαντικά πρακτικά προσκόμματα και τις ουσιαστικές αλλαγές για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά χρειάζεται αναθεώρηση του κανονισμού και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταφέρουμε αυτό διότι ε, ξεκίνησε μια διεξοδική διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού του 2015 την αμεδίκονουσε όσους είχαν εκφράσει την άποψή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διοργανωτές προηγούμενων πρωτοβουλίων και πάνω από 5.000 άτομα απάντησαν στη δημόσια διαβούλευσή μα. Εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνατε μια πολύ σημαντική συνεισφορά και στο ψήφισμα του 2015 και στα όσα έγιναν εν ώψη ε, του ψηφίσματος ιδίας πρωτοβουλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σέπφλιν και τους υπόλοιπους εισηγητές τον κύριο Βαλέσα, τον ε, κύριο Τζαμπάσκι για τα όσα έκαναν. Και επίσης ε, θα δείτε αν εξετάσετε την πρότασή μας ότι οφείλουμε πολλά στα όσα έγιναν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή σύντομα. Η αναθεώρηση τη διαδικασία τα τελευταία ένα-δύο χρόνια μα οδήγησε σε πολύ σαφή συμπεράσματα για το ποια είναι τα προβλήματα και πώ μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό ακριβώ και υποβάλλουμε την πρότασή μας, υποβάλαμε την πρότασή μα στι 13 Σεπτεμβρίου. Οι νέοι κανόνε που προτείνουμε ε, σημαίνουν ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να προτείνει κάποιο και να υποστηρίξει πρωτοβουλίε. Θα μπορούν να τύχουν μεγαλύτερη υποστήριξη και οι διοργανωτέ μπορούν να έχουν και ένα κεντρικό σύστημα για διαδικτυακή συλλογή υπογραφών, το οποίο θα διαχειρίζεται πλήρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαδικασία υπογραφή θα είναι απλοποιημένη και οι πολίτε θα μπορούν να υπογράψουν και μέσω ηλεκτρονική ε, ταυτότητα. Θέλουμε να ε, αντιμετωπίσουμε και ένα σημαντικό κενό, το οποίο δεν έχει επιληθεί μέχρι τώρα. Επειδή υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε απαιτήσει των κρατών μελών, υπάρχουν ακόμα πολίτε που δεν μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. Με τους νέους κανόνες προτείνουμε όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών, ανεξάρτητα από το που διαμένουν, να μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Μειώνοντας ε, την ελάχιστη ηλικία στα 16 έτη επίσης, ε, κάνουμε μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Νεολαία να συμμετέχει και να εισακουστεί η φωνή της, να μας προτείνει τις ιδέες της και να μάθουμε τι είναι αυτό που του ενδιαφέρει. Έτσι θα έχουμε 10 εκατομμύρια επιπλέον νέους Ευρωπαίους να μπορούν να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες. Μπορεί οι millennials να μην μπορούν να ψηφίσουν στα περισσότερα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να εισακούγεται η φωνή τους και έχουν πολλά να συνεισφέρουν στο ευρωπαϊκό όραμα. Ε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ναι δεν είναι μια γενιά η οποία έχει ιδεολογία αλλά είναι ιδεαλιστές και πιστεύω ότι αυτά ε, θα πρέπει να αναφέρονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία παρακολούθηση. όταν μια πρωτοβουλία καταφέρει να επιτύχει την υποστήριξη του ενό εκατομμύριου υπογραφών. Από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ελεύθερη να αποφασίσει κατά πόσον θα δώσει συνέχεια, αλλά πριν αντλήσει τα συμπεράσματά τη, θα πρέπει να γίνει ουσιαστική συζήτηση και δέσμευση από όλα τα θεσμικά όργανα και τα συμβουλευτικά όργανα που μπορούν να διαδραματίσουν και αυτά το ρόλο του. Ε, σε ε, ε, επίπεδο βεβαίως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στην κοινοβουλευτική, στη συμμετοχική δημοκρατία, μπλουτίζει την κοινοβουλευτική δημοκρασία και τη συμπληρώνει και νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στην ευρωπαϊκή πολιτική και στη χάραξη πολιτική. Μπορεί να βελτιώσει τα όσα κάνουν οι πολίτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βοηθά τη δημοκρατική ε, διαδικασία πέραν των συνόρων ε, και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προωθεί ιδέες που πολλοί πολίτες ενδιαφέρονται, για τις οποίες πολλοί πολίτες ενδιαφέρονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για όλους εμάς αυτό το συμμετοχικό εργαλείο να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αποτολιτών, ε, εάν μπορεί να ε, χρησιμοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, θα είναι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε αποτελέσματα πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές για να μπορέσουμε να δείξουμε και αυτά αποτελέσματα πριν τις εκλογές. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε τον εισηγητή της Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων, τον κύριο Σέπφλιν. Θα σας δώσω το λόγο για τρία λεπτά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας επισκέπτεστε σήμερα το απόγευμα. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για αυτή την περιγραφή που κάνατε και Έχω να διαφωνήσω μόνο μαζί σας σε ένα σημείο επί της αρχής. Είπατε πως ο πλουραλισμός είναι η καρδιά της δημοκρατίας. Εγώ θα έλεγα πως είναι η διακυβέρνηση μέσω ε, συγκατάθεσης. Ε, νομίζω ότι μπορεί να μην έχει συνέπειες για τα όσα θα πούμε σήμερα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε πως δεν δεχόμαστε όλοι πως ο πλουραλισμός είναι η καρδιά της δημοκρατίας. Να πω και δύο λόγια για το γεγονός πως η συμμετοχική δημοκρατία δεν είναι άμεση δημοκρατία. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Και ίσως δεν το κατανοούν όλοι εδώ πως όλα λειτουργούν αρκετά καλά στην Λετωνία και στη Φιλανδία και νομίζω είναι μοναδικές δύο χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ε, τέτοιου είδους παράλληλο εργαλείο, Α, όχι όμως και για τους υπόλοιπους. Η βασική δυσκολία στην οποία αναφερθήκατε και εσείς, το άρθρο 11, είναι αυτό το invite. Δηλαδή καλούμε. Το πρόβλημα για μένα είναι το ότι αν καλέσουμε κάποιο, απλώ του απευθύνουμε μία πρόσκληση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σκεφτεί ε, σοβαρά ε, τι γίνεται με το μονοπόλιο της πρωτοβουλίας που έχει. Για την ομοθεσία πρέπει να σου πω πως αυτό βρίσκεται στην καρδιά του τρόπου με τον οποίο έχουν δομηθεί τα θεσμικά όργανα. Και η προσωπική μου σκέψη είναι ε, πως θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο είδους ε, ε, αρχή ε, η οποία θα επιτρέπει να αποφασίζουμε σε κάθε περίπτωση εάν χρειάζεται νομοθεσία ή όχι. Αυτές οι ίδιες πρωτοβουλίες που είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση της γλυφωσάτης και τα Λυπάσματα. Αυτή είναι πραγματικά ένα καλό παράδειγμα. Υπάρχουν κανένα δύο ακόμα, είπατε, μας είπατε, μπορείτε θα μας δώσετε συγκεκριμένε πληροφορίες. Τώρα για την διαβούλευση, ε, τη δημόσια διαβούλευση που έληξε στις 16 Αυγούστου. Θα θυμόσαστε κι εσείς τη δήλωση που είχατε υποβάλει την Άνοιξη που είπατε πως θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου αυτή η πρωτοβουλία πολιτών ε, οπότε η διαβούλευση δεν έτρεξε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Εσείς ε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση που προσπαθείτε να επανασχεδιάσετε τον ολόκληρο μηχανισμό, αλλά δεν ξέρω σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών αν του έχουμε δώσει ε, αρκετό χρόνο. Τώρα για την ηλικία των 16 δεν μπορώ να πω ότι είμαι κατά επί της αρχής, αλλά θα πρέπει να ξέρετε πως το μεγάλο βάρος αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι η 65 και πάνω και δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο προσωπικά στον εαυτό μου ίσως βέβαια ως εκπροσωπώ ένα αριθμό από αυτούς αλλά λαμβάνοντας υπόψη ε, το ότι όλοι λέμε τα νιάτα είναι καταπληκτικά αλλά νομίζω ότι η δημοκρατία είναι να έχουν ένα αποφασιστικό ρόλο και πάνω των 65. Γιατί οι σημερινοί νέοι θα ζήσουν μέχρι τα 130. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να λάβουμε υπόψη και τι ηλικίε στις οποίε αναφέρομαι οποιαδήποτε σώρευση εξουσίας, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς εξασφαλίζουμε πως οι αρμοδιότητες αυτές δεν θα τις καταστραχθεί αυτούς που έχουμε. Γιατί ξέρετε πως υπάρχει πάντα το σχετικό νομικό θέμα του ποιος φυλάει τους φύλακες. Πού είναι οι θεσμοί της ε, δημοκρατικής λογοθεσίας. Πολλές αρμοδιότητες που πολύ εξορθολογισμένα έχετε παρουσιάσει εσείς, αλλά λογοδοσία λογοδοσία. Σας παρακαλώ πολύ μπορείτε να πείτε δύο λόγια. Και λυπάμαι που ξεπέρασα τον χρόνο μου, συνήθως δεν το κάνω, αλλά είχα πολλά να πω. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαλέντσα βρίσκεται εδώ από την Επιτροπή Αναφορών και είσαστε εισηγητής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στο άρθρο 14 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να είναι πιο ισορροπημένες οι, ακρο... ακροάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες ε, Πολιτών, ε, ώστε, να εκπροσωπούνται, ώστε να εκπροσωπείται ευρύ φάσμα θέσεων. Ενώ λοιπόν ε, θέλετε μια πιο συμμετοχική προσέγγιση και η οποία εγκρίνεται και από τον Ευρωπαίο Διαμισολαβητή, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Και όσον αφορά το άρθρο 15 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να παρατείνει την προθεσμία για απάντηση από 3 σε πέντε μήνες. Δεδομένου του χαμηλού αριθμού επιτυχημένων πρωτοβουλειών πολιτών μέχρι στιγμής, διότι ελάχιστες ε, έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένες ε, δράσεις από πλευράς της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προβλέπει τις αντιδράσεις σε, σε μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτών. Και όσον αφορά το άρθρο 16 και την ε, πρόταση για ε, οικονομική ενίσχυση προς τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο επικροτούμε, αλλά και πάλι στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί η διάταξη αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καλέσει και τον εισηγητή, του συντάκτη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού. Αναρωτιέμαι αν είναι παρόν ο κύριος Τζαμπάσκι. Δεν νομίζω ότι είναι παρόν. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στους κοιόδης εισηγητές, ε, ξεκινώντας από την ΑΦΚΟ. Την κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τίμερμανς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να εξετάσουμε μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για να πετύχουμε περισσότερη συμμετοχή των πολιτών μας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και ως ε, ε, πρώην μέλος της Συνταγματικής Συνέλευσης ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που προβλέπεται ε, ελάχιστη, ενιαία ελάχιστη ηλικία 16 ετών. Ε, επί πολλά χρόνια αγωνίζομαι γι' αυτό. Και άσχετα από τις ε, δημογραφικές εξελίξεις υπάρχουν εκατομμύρια νέων ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν την Ευρώπη. Και σε όλες ε, τις ε, συζητήσεις μας νομίζω θα πρέπει να λαμβάνετε αυτό υπόψη. Επίσης ε, βρίσκω ότι είναι πολύ καλό το ότι προβλέπετε την καταχώρηση των πρωτοβουλειών, την δυνατότητα με, υποστήριξης για τη μετάφραση και πολλές άλλες προτάσεις τις οποίες ε, υποστηρίζω όλες. Νομίζω ότι το σχέδιο του κειμένου ακολουθεί την σωστή κατεύθυνση. Τρεις παρατηρήσεις ε, θα ήθελα να κάνω, τρεις ανησυχίες έχω. Καταρχάς, ε, τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να διαδώσουμε περισσότερο τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, διότι διαπιστώνουμε ότι πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν τι δικαίωμα έχουν. Δεύτερον, ίσως θα έπρεπε πάλι από κοινού να σκεφτούμε ε, πώς μπορούμε να στηρίξουμε οικονομικά τις πρωτοβουλίες, για παράδειγμα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως είναι η Ευρώπη για τους πολίτες ή το, πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και ε, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και δεν ξέρω μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς, διότι όσον αφορά την ενιαία διαδικασία για ε, που προτείνεται εμένα μου φαίνεται πολύ πιο πολύπλοκη από πριν, ε, αλλά μήπως πρέπει να διαβάζω πιο προσεκτικά το κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ο Σαλ Γκέρενς. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω την πρόοδο που μας ανέφερε ο κύριος Τίμερμενς για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, ιδίω όσον αφορά την εξέλιξη της ε, συλλογής υπογραφών διαδικτυακά, την ε, μερική αποδοχή των πρωτοβουλειών, την ευελιξία όσον αφορά την ημερομηνία από την οποία ισχύει η διάρκεια των 12 μηνών ε, της συλλογής των υπογραφών και η μετάφραση της πρωτοβουλίας σε όλες τις επίσημες ε, γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μέτρα τα οποία ε, στόχο έχουν να βελτιώσουν το σύστημα και να το κάνουν πιο δημοφιλές ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχω παρόλα αυτά κάποιες ερωτήσεις, περισσότερο σε επίπεδο κατανόησης και να έχω να κάνω και μια πρόταση. Όσον αφορά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων, Υπάρχουν δύο συστήματα, αν κατάλαβα καλά ε, το σημείωμά ε, ε, Δύο συστήματα τα οποία μπορεί να συνεπάρχουν. Ένα πρώτο σύστημα το οποίο ε, προβλέπει ότι δίνεται όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως και διεύθυνση και ένα δεύτερο όνομα, επώνυμο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία της ταυτότητάς του. Το θέμα το οποίο θα ήθελα να σήξω δεν είναι κεφαλαιόδου σημασία μεν, αλλά δημιουργεί κάποια ερωτηματικά τι γίνεται όταν κάποιος έχει διπλή ηθαγένεια. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάποιος να μπορεί να υπογράψει δύο φορές. Ε, εντάξει, δεν θα συμβεί ε, χιλιάδες φορές, αλλά επειδή ακριβώς ε, επικαλούμαστε και τις δυσκολίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν, σας θέτω και το συγκεκριμένο ερώτημα. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω και μία πρόταση που έχει γίνει ήδη στα πλαίσια της συζήτησης για την έκθεση του κυρίου Σέπφλιν. Ε, η πρώτη αφορά την μερική εγγραφή που επιτρέπεται ε, βάσει της πρότασής σας. Το δεύτερο είναι να γνωρίσουμε τι γίνεται με το σκέλος το οποίο δεν θα ε, λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μας η πρόταση ε, περιλάμβανε συνέχεια αυτού του σκέλους από τις αρμόδιες αρχές είτε ευρωπαϊκές είτε σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Ε, κατά την άποψή μας αυτό αποτελεί ε, καλή διοικητική πρακτική η οποία υπάρχει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και ε, δεύτερον κάτι το οποίο θίξατε στη διάρκεια της συζήτησης για την έκθεση Σέμφλιν και υποβάλαμε και σχετική τροπολογία για το ενδεχόμενο οι πολίτες να προτείνουν επίσης και κάποιες τροπολογίες, τροποποίησεις δηλαδή, στο πρωτογενές δίκαιο διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προτείνει και αλλαγές ε, των συνθήκων και τροπολογίες. Θα θέλαμε και οι πολίτες ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών να κάνουν τέτοιες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εύστοχη παρατήρηση. Ο κύριος Τερικάμπρας από τους Πρασίνους τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς να σας πω πως αυτή η πρωτοβουλία είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για τη συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη τα σοβαρά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρόλο που συμπεριλαμβάνει κάποια από τα αιτήματα των εμπλεκομένων, κατά τη γνώμη μας δεν επαρκεί για τρία βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρωτοβουλίας. Γιατί εσείς λέτε πως θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή αν η πρωτοβουλία αυτή κτλ. κτλ. Όμως η διατύπωση αυτά δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε ε, να ανατρέψει την απόφασή της να μην καταχωρήσει μια πρωτοβουλία λόγω ε, πολλών προβλημάτων ε, λόγω δηλαδή του Μανόρτσεφ, για παράδειγμα, και κάποιων άλλων θεμάτων. Και επίσης, το γεγονός πως χρειάζεται νομική καταχώρηση αυτής της πρωτοβουλίας και αυτό αποτελεί πρόσκομα. Γιατί εσείς είσαστε και δικαστής και διάδικος στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο θα κάνει την εξέταση, την νομική για την καταχώρηση αυτής της πρωτοβουλίας. Μετά η συνέχεια, το follow-up. Είναι επίσης σημαντικό και είναι ουσιαστικό για να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε το κατάλληλο follow-up και όχι απλώς να απευθύνουμε μια πρόσκληση όπως είπε και ο συνάδελφος και ο Σόπφλιν. Διαφορετικά είναι ένα εργαλείο άχρηστο και το μόνο που θα δημιουργήσουμε είναι εκνευρισμό. Κάτι το οποίο δεν είναι χρήσιμο. Παρόλο που είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Περιμένουμε λοιπόν πιο ε, τεκμηριωμένη εξήγηση στην περίπτωση που δεν λαμβάνει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν δεν λαμβάνει δράση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και νομίζω ότι Παράλληλα, αν δεν σας πειράζει κύριε Τίμερμανς, θα συνεχίσουμε με τους σκιώδεις της Επιτροπής Αναφορών έτσι ώστε να απαντήσετε ε, στα θέματα που αφορούν και τις δύο επιτροπές. Η κυρία Μίτση. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς χαιρετίζουμε αυτή την ε, αναθεώρηση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία πραγματικά καθυστέρησε, γιατί η αρχική μορφή απογοήτευσε τους πολίτες μετά τις πρώτες υποσχέσεις που είχε δώσει. Εγώ έκανα μια γρήγορη ανάγνωση και πρέπει να σας πω πως υπάρχουν εξή σημεία στα οποία θέλω να σταθώ. Ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών, για παράδειγμα. 800.000 υπογραφές. Γιατί όχι ένα εκατομμύριο τι θα γίνει. Ε, αν είναι 800.000 και όχι ένα εκατομμύριο, θα τα πετάξετε, θα τα αφήσετε στην άκρη. Επίση, υπογραφέ να μετριούνται στα κράτη-μέλη. Και τι θα γίνει. Αν ένα πολίτη ζει σε ένα κράτο μέλο, όπου δεν είναι το κράτο υπηκότητα, Πώς θα τον αντιμετωπίσετε. Επίση. Χαιρετίζω το νέο άρθρο για την ενημέρωση και την ε, βοήθεια που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους οργανωτές των πρωτοβουλειών, αλλά θέλουμε να ε, περιγράφεται ε, πιο σαφώς τι είδους αρρωγή θα προσφέρεται, για παράδειγμα, η ενημέρωση. Τώρα για την ομάδα οργανωτών, εδώ θα αντιμετωπίσουμε και την περίπτωση νομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ομάδες για παράδειγμα παράγραφος 5 και 6 για την ευθύνη και τις κυρώσεις επί των οργανωτών, ε, πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάτι αντίστοιχο και να δούμε και πώς θα επηρεάσει τις πρωτοβουλίες. Επίσης, κάτι το οποίο θα δώσει οργανωτές την ευελιξία του πότε θα ξεκινάει η συλλογή υπογραφών. Αυτό είναι καλοδεχούμενο, αλλά τι επίπτωση θα έχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίζει ε, και τι θα γίνει αν έχουμε μονομερική καταχώρηση. Χαίρομαι πως έχουμε αυτή τη νέα ε, δυνατότητα της online καταχώρησης υπογραφών ε, αλλά να με εξηγήσετε πώς θα λειτουργήσει, πόσο απλουστευμένο και αναρμονισμένο θα είναι. Αλλά νομίζω ότι οι ανησυχίες βασίζονται στο ότι δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματική θα είναι η συμμετοχή μέσω των υπογραφών. Δηλαδή, πώς ακριβώς θα το διαχειριστούμε και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δίνει σάκα και οστά σε αυτά που επιθυμούν οι πολίτες. Γιατί είναι μια πραγματικά ε, βαριά προσπάθεια. Thank you very much and I would... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την πληροφορία που μόλις έλαβα από την Τανούτα Χίπνερ. Εκλήθη να συμμετάσχει σε μια πολύ επίγουσα συνάντηση για ένα πάρα πολύ επίγον πολιτικό θέμα. Μπορείτε λοιπόν να περάσετε το απόγευμά σας μαντεύοντας ε, ποιο είναι αυτό το θέμα. Πάντω ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρούσα και σε εσά κύριε Τίμερμαν και στις δύο επιτροπές μας. Και μας ε, έχει στείλει και κάτι εικονίδια και λουλουδάκια στο μήνυμα, στο κινητό. Ε, ζητά λοιπόν ταπεινά συγγνώμη. Ας συνεχίσουμε. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Δύο λεπτά το πολύ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, το δικαίωμα πρωτοβουλίας, ε, αυτό που ονομάζεται Citizens Initiative, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ενισχύει τα στοιχεία συμμετοχικής δημοκρατίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως πρέπει να κοιτάμε την πολιτική ουσία καταρχάς και όχι τον τύπο. Δηλαδή πρέπει να βρούμε προϋποθέσεις οι οποίες να βοηθούν τους πολίτες να συμμετέχουν και αυτό έχει σχέση και με τον τρόπο συλλογής υπογραφών και με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται. Και φυσικά όσο πιο απλό είναι το σύστημα, τόσο πιο σημαντική είναι η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν ο πρώτος στόχος να απλοποιήσουμε τη διαδικασία νομίζω ότι πρέπει να υπηρετηθεί από αυτή τη νέα πρόταση που κατεβάζει η Κομισιόν. Είδαμε τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν και θεωρώ ότι με τις προτάσεις που διαμορφώνονται και τις ερωτήσεις θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα πιο απλό για να μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική την πρωτοβουλία των πολιτών. Υπάρχει όμως ένα θέμα ουσίας κύριε Τίμερμανς και αυτό έχει σχέση με τη διαδικασία κατά την οποία η Κομισιόν ελέγχει τις νομικές προϋποθέσεις, κατά πόσο δηλαδή τυπικά είναι ορθή η πρόταση που υποβάλλουν οι πολίτες. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει η Κομισιόν. Αυτό πρέπει να το κάνει ένα άλλο όργανο το οποίο θα δει ποιες είναι οι νομικές προϋποθέσεις και θα δεχθεί ή θα απορρίψει την αίτηση των πολιτών. Προτείνω λοιπόν, επειδή κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το κάνει ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί δικιά του διαδικασία και μπορεί να καλέσει για νομοθετική πρωτοβουλία την Κομισιόν, να είναι μια αρμοδιότητα που να δώσουμε στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή ο οποίος θα μπορούσε να εξετάσει τις τυπικές προϋποθέσεις και αν θεωρεί ότι αυτές υπάρχουν, τότε να στέλνει την πρόταση στην Κομισιόν, η οποία βεβαίως στη συνέχεια θα πρέπει να συναντηθεί με τους πολίτες για να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα ασκηθεί η νομοθετική πρωτοβουλία. Διότι διαφορετικά η Κομισιόν θα είναι αυτή που ελέγχει τις νομικές προϋποθέσεις, αλλά είναι ταυτόχρονα και αυτή που θα αναγκαστεί να προχωρήσει στην νομοθετική πρωτοβουλία. Και αυτή, αυτό δημιουργεί μια σύγκρουση συμφερόντων που νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την άρουμε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων δίνοντας τις εξουσίες ελέγχου της, νομ, της νομικής πληρότητας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Now the floor goes to Mrs. Το λόγο έχει η κυρία Πεσέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κύριε Τίμενας που ήρθατε και πάλι να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τους πολίτες. Εγώ ήμουν εισηγήτρια μαζί με τον κύριο Σέπφλιν σε μια προηγούμενη έκθεση για το θέμα αυτό και μου αρέσει που μιλάμε για τον πυρήνα της δημοκρατίας εδώ και για το ότι ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις, αν είναι η συνένεση, αν είναι ο πλουραλωματισμός, πλουραλισμός. Εγώ νομίζω θα πρέπει να είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή ε, και στην νομοθεσία αλλά και μέσω εκλογή ερετών. Με τον τρόπο αυτό οι ευρωπαϊκοί ε, ε, πολίτες μπορούν να νομοθετήσουν. Το λέμε πρωτοβουλία, αλλά ουσιαστικά η πρωτοβουλία έχει ένα σκοπό και δεν μπορεί να έχει το μονοπόλιο αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το εργαλείο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε ξεδιπλώσει επαρκώς Όλη αυτή η διαδικασία νομίζω κατάφερε να εντοπίσει ποια είναι τα βασικά προβλήματα και το πρόβλημα ήταν ότι είχαμε απορρίψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προτάσεων. Το, πολύ λίγες πρωτοβουλίες φτάνουν ε, να καταλήξουν και το γεγονός πως περνάμε ε, μια διαδικασία η οποία τρέχει παράλληλα με αυτήν την έκθεση για τον ευρωπαϊκό πολίτη και για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Οπότε καταλαβαίνετε στα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και στοιχεία από το εργαλείο της πρωτοβουλίας. Θέλω να πω κάτι το οποίο είχαμε και στην προηγούμενη έκθεση συνενετικά και στη φετινή. Γιατί δεν καταφέρνουμε αυτό το μεγάλο ε, ε, νούμερο των υπαλλήλων και ε, εξοπλισμού που έχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλα τα γραφεία ε, του Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα να, λειτουργήσουν, στην Ευρώπη με συγχωρείτε, να, να λειτουργήσουν ως μια ενιαία θηρίδα και μέσω αυτών να φτάνουν οι πληροφορίες σε εμάς. Νομίζω ότι θα ήταν ένας τρόπος αυτός να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία Πολιτών. Και τώρα ε, για να μετρήσουμε τα νούμερα. Χρειαζόμαστε να λάβουμε υπόψη τι είπε το ελεκτικό συνέδριο και θα πρέπει για παράδειγμα να δούμε την πρόσφατη και αρνητική ε, απόφαση του ελεκτικού συνέδριου σχετικά με το θέμα που συζητάμε. One more. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρούσα είναι και η κυρία Εύη από την Επιτροπή μου, αλλά δεν είδα να ζητάτε το λόγο. Θέλετε το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Τίμερμανς, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς είπατε ότι θέλετε να δώσετε συνέχεια στην πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών για να σταματήσει η γλυφοσάτη και το δικαίωμα στο νερό στην αρχή της παρέμβασής σας. Πώς συνάδει αυτό με την απόφαση που λάβατε τη Δευτέρα για την ανανέωση της ε, άδειες κυκλοφορίας αυτή τη ουσίας. Ε, διαπιστώνω κάποια συνέπεια στα όσα λέτε σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Ανανεώνεται η άδεια μιας ουσίας η οποία είναι πιθανόν ε, καρκινογόνος και τοξική για το οικοσύστημα. Όσον αφορά την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, ένα τόσο σημαντικό ε, εργαλείο το οποίο δυστυχώς απογοήτευσε πάρα πολλούς πολίτες μέχρι σήμερα που πίστεψαν σε αυτό το εργαλείο και δυστυχώς τους πλήγωσε η πλήρης αδράνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που δεν ανταποκρίθηκε στους προβληματισμούς των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να σας ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις λοιπόν για αυτή τη νέα πρόταση όσον αφορά το παραδεχτό των προτάσεων των Ευρωπαίων πολιτών που αφορούν τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, τα όσα συνέβησαν με την πρωτοβουλία Stop TTIP, η οποία αρχικώς ε, θεωρήθηκε μη παραδεκτή ακριβώς ε, γιατί αφορούσε προπαρασκευαστικές πράξεις. Ε, γιατί δεν ε, διευκρινίζεται καλύτερα αυτή την πτυχή στη νέα πρόταση. Επίσης, εσείς είπατε ότι για να ενισχύσουμε τη δημοκρατική αρχή και τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα μπορούσε να γίνει δεκτή μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που προβλέπει και αλλαγή των συνθήκων ώστε να συμμετέχουν πραγματικά οι πολίτες στις διαδικασίες αυτής της Ευρώπης. Ε, και μία ακόμα ερώτηση όσον αφορά ε, την αιτιολόγηση σε περίπτωση απορριψη ε, μιας πρότασης, όπως συνέβη για παράδειγμα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το Minority Safe Pack. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη διατύπωση για τις σημαντικές αυτές πτυχές για να μπορέσει κάποιος να αποδεχτεί ή να απορρίψει μία πρόταση ε, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ε, και εσείς είστε η τελευταία ομιλήτρια από πλευράς ε, ε, σκιωδών εισηγητών, αλλά έχω και άλλα τέσσερα μέλη που θέλουν να λάβουν το λόγο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σκιώδεις εισηγητές. Ε, ο πιο λογικός τρόπος λοιπόν είναι να δώσουμε το λόγο και σε αυτούς και μετά να απαντήσετε στη συνέχεια κύριε Τίμερμαν. Συμφωνείτε? Ωραία. Ο κύριος Δουρά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί βέβαια θα πρέπει να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε μας για τις προτάσεις σας γιατί όπως είδα ε, σεβαστήκατε την υπόσχεσή σας και ήρθατε να μας τα παρουσιάσετε. Γι' αυτό σας ευχαριστώ και για το ουσιαστικό της συζήτησης. Νομίζω ότι γενικά το κείμενο είναι βελτιωμένο. Εκεί δεν έχω πρόβλημα. Όμως έχω μια ερώτηση για το αν πιστεύετε πραγματικά πως είναι μόνο βελτιώσεις λειτουργικές, ηλικιακό κτλ. που θα βοηθήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες να αισθανθούν ότι και πάλι τους αφορά αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Γιατί εντάξει, οι πλατφόρμες αυτές σε όλες τις γλώσσες λοιπά πολύ καλά. Αλλά μήπως υπάρχει και πολιτικό πρόβλημα και μήπως το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα δεν είναι μόνο αν θα μπορούμε και για την κατάργηση, για παράδειγμα, για την τροποποίηση να έχουμε μια πρωτοβουλία και όχι μόνο για αυτό που ήταν στο παρελθόν, αλλά για το γεγονό πω δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα, Πώ δεν έχουμε εξηγήσει, εσεί μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ότι δίνεται κάποια συνέχεια σε μια απόρριψη, σε μια αποδοχή πρωτοβουλία. Γιατί Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει να μπορεί μέσω ψηφίσματος ε, να δώσει τη δυνατότητα να συζητηθεί ένα θέμα που αφορά ε, μέσω πρωτοβουλία στους Ευρωπαίους πολίτες και μέσω αυτής της συζήτησης ενδεχομένως να το μετατρέψει και σε νομοθετική πρωτοβουλία. Μήπως λοιπόν δεν μπορούμε να βελτιώσουμε και το πολιτικό περίβλημα αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και να μην δούμε μόνο τις πρακτικές πτυχές οι οποίες βέβαια και αυτές όπως σας είπα εδώ είναι βελτιωμένες. Ευχαριστώ πολύ. Nice to see you in this committee also. Ε, θα μιλήσω πολωνικά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, είμαι οπαδός της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και επικροτώ τις τροποποίησεις αυτές. Τρεις ερωτήσεις έχω, αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, Κάθε πολίτης ε, που συμμετέχει σε μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει την, την πεποίθηση ότι η διαλειτουργικότητα, οι, ηλεκτρονικές υπογραφές ε, και λοιπά θα διασφαλίζονται όσον αφορά τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Πρέπει οι πολίτες να ε, έχουν εμπιστοσύνη όσον αφορά τις πτυχές προστασίας των δεδομένων. Εάν δεν προωθηθεί σωστά η πρωτοβουλία αυτή, θα είναι άλλη μια πρωτοβουλία που θα πέσει στο κενό. Θα πρέπει λοιπόν να τη διαφημίσουμε. Επίσης, μιλάμε για πρωτοβουλίες διασυνοριακές. δεν θα πρέπει να επανέλθουμε στη συζήτηση σχετικά με διασυνοριακούς οργανισμούς και ιδρύματα. Δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις διασυνοριακές πρωτοβουλίες πολιτών το 2002, το 2014 είχαμε τη συζήτηση αυτή, δεν καταλήξαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Μήπως θα μπορούσαμε να την επαναλάβουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζέμις, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμανς, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και ίσως να σας εκπλήσει ότι στηρίζω οτιδήποτε ε, βοηθήσει να ε, έχουμε δημοκρατία με νόημα στα θεσμικά όργανα και μέχρι ε, το Brexit. Μου φαίνονται πολύ λογικά όλα αυτά που ακούω. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως έχουν, υπήρξαν μέχρι τώρα 60 τέτοιες πρωτοβουλίες και ενώ κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο μέλλον και τους νέους ανθρώπους λέγοντας ότι οι προτινόμενες τροποποίησεις αυτούς θα βοηθήσουν. Μήπως ε, θα μπορούσατε να ξανακοιτάξετε τις προηγούμενες 60, συγκεκριμένα τις 54 που απορρίφθηκαν, ε, για να δούμε μήπως υπάρχουν ε, πράγματα που μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πούν ότι ακούστηκε η φωνή μου, εξετάστηκε το θέμα και έχουμε αυτά αποτελέσματα. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, οι Ευρωπαϊκέ Πρωτοβουλίε Πολιτών ε, θα είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Υπάρχει τρόπος να γίνουν κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να υπάρχει ε, μια μέση οδό ώστε να έχουν περισσότερη υπεποίθηση οι πολίτες. Και επίσης, αντί να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, μήπως μπορούμε να μιλάμε για Πρωτοβουλία Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το λέω αυτό, διότι εδώ μιλάμε συνέχεια για περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αυτό θέλουμε να πετύχουμε, τότε θα πρέπει ε, ακριβώς αυτό να μπορούν να επικαλεστούν οι πολίτε, ότι είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πέτερ Γιάρ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα που είδα προς το τέλος μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Όλα είχαν πάει λίγο πολύ καλά, οι πολίτες βρέθηκαν εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, κατόπιν όμως ε, εγκατέλειψαν απογοητευμένοι τις Βρυξέλλες. Ε, μπορεί να μην είναι θέμα νόμων ή πολιτικής βούλησης. Ε, υπευλήθη η πρωτοβουλία των πολιτών. Ωραία, οργανώνουμε ακροάσεις. Ε, διαπιστώνουμε ότι μπορεί να είναι αιτιολογημένη η πρωτοβουλία σας, ε, αλλά μπορεί να να αντίκειται στους νόμους, να μην, να μην έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία για κάτι τέτοιο. Οι πολίτες ε, λοιπόν ε, περήφανοι που ε, καταφέρανε να φτάσουν μέχρι εκεί έρχονται στις Βρυξέλλες αλλά επιστρέφουν στις πατρίδες τους απογοητευμένοι. Πώς μπορούμε όπως είπε και η συνάδελφος να κάνουμε πιο δεσμευτικές τις πρωτοβουλίες πολιτών. ώστε τουλάχιστον να οδηγήσουν σε πολιτική δράση οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών πρωτοβουλία των πολιτών, δράση των πολιτών, προσέλευση στις Βρυξέλλες, αλλά θα πρέπει κάτι να γίνει μετά από αυτό. Δεν μπορούμε να του πούμε ότι οι Βρυξέλλες έχουν δικό τους θεματολόγιο. Η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, λοιπόν, ε, πώς μπορούν να ενεργήσουν. Έχετε κάποια ιδέα πέρα από την νομοθεσία. Να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους ε, όσοι συμβάλλατε με σημαντικές ερωτήσεις. Ε, δίνω λοιπόν ε, προς τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε σε κάποια από τα θέματα αυτά, ενώ άλλα είμαι σίγουρη ότι θα τα απαντήσετε αυτό το χρόνο στις επιμέρους επιτροπές. Ο κύριος Τίμερμαν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις. Τις υπόλοιπες ε, θα τις απαντήσουμε γραπτώς. Οι συνεργάτες μου έχουν καταγράψει τις ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές είναι πολύπλοκες. Ε, δεν είναι λοιπόν έλλειψη σεβασμού. Έλλειψη γνώσεων είναι, αν δεν καταφέρω να απαντήσω σε όλες. Αλλά θα φροντίσω να απαντήσουμε σε όλες τελικά. Δεν ε, θα ξεκινήσω συζήτηση με τον κύριο Σεφλίν με όλο το σεβασμό για τη φύση της δημοκρατίας και για το... Ε, ε, βασίζεται στη συγκατάθεση ή αν έχει να παίξει ρόλο και η διαφοροποίηση αλλά στην ευρωπαϊκή μας δημοκρατία Ε, το πόσο καλή είναι η απόφαση το, της πλειοψηφίας ε, εξαρτάται από το πόσο σέβεται τη μειοψηφία, διότι η σημερινή πλειοψηφία αύριο θα είναι μια μειοψηφία. Και αν ε, κοιτάξετε την Ευρώπη σε υπηρετική κλίμακα, αν την δείτε ως Ήπειρο, όλοι μειονότητα είμαστε. Δεν υπάρχει κάποια δεσπόζουσα πλειοψηφία, πλειονοτική ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λειτουργεί η Ευρώπη και έτσι λειτουργεί επιτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ικανοποιήσω και την κυρία James. Εκεί έγκυται η επιτυχία της και πιστεύω ότι όσο περισσότερο σέβεται κανείς την μειοψηφία, τόσο περισσότερο σεβασμό συγκεντρώνει και η πλειοψηφία όσον αφορά την ε, ευχέρειά της ε, να κάνει αυτό που θέλει. Ο κύριος Σεφλίν ε, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν πρόκειται για εργαλείο άμεσης δημοκρατίας, πρόκειται για διαβούλευση η οποία μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να οδηγήσει στην υιοθέτηση νέας νομοθεσίας από τους συνομοθέτες. τους πολλούς από εσά ε, που θεωρούν ότι αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό βήμα πρόοδου αλλά που θέλουν να προχωρήσουν πιο πέρα, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε πέρα από ό,τι μας επιτρέπει η συνθήκη. Και όσο λυπηρό και να φαίνεται αυτό από μια συγκεκριμένη ε, άποψη, Δεν μπορούμε να δώσουμε δικαίωμα πρωτοβουλίας στους πολίτες που να απαγορεύεται από τη συνθήκη και που να μην έχει καν το κοινοβούλιο. Η Επιτροπή είναι θεματοφύλακας των συνθήκων αλλά και των δικαιωμάτων που αποκτά μέσα από τη συνθήκη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρωτοβουλίας. Τούτου λεχθέντος ε, πιστεύω ότι εάν υπάρχει το εργαλείο της ε, πρωτοβουλίας πολιτών έχει κανείς τουλάχιστον την πολιτική υποχρέωση να αιτιολογήσει ε, την αντίδρασή της. Εφόσον η πρωτοβουλία των πολιτών ε, συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό υπογραφών που είναι απαραίτητες. Πρέπει δηλαδή να αιτιολογήσει κανείς την αντίδρασή του ε, ακόμα και εάν δεν οδηγηθεί σε νέα νομοθεσία. Ε, δεν είμαι βέβαιος αν αυτό ζητά ο κύριος Σεφλίν, αλλά αυτό είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει. Ο κύριος Σεφλίν αντιστρέφει το επιχείρημα. Λέει ότι πρέπει να αιτιολογήσει κανείς για, σε περίπτωση που δεν νομοθετήσει. Δηλαδή, νομοθεσία εκτός εάν υπάρξει σωστή αιτιολόγηση. Νομίζω ότι αυτό όμως ε, είναι μάλλον υπερβολικό. Συμφωνώ όμως ε, ότι θα πρέπει ε, να είναι επαρκώς αιτιολογημένη η αντίδραση. Επίσης, άκουσα ευρωβουλευτές να επιχειρηματολογούν ότι η καταχώρηση δεν πρέπει να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έχει να κάνει και με τις νομικές της υποχρεώσεις. Ε, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ε, ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, θα, θα παρέμβει το... Θα επέμβει το δικαστήριο και αυτό έχει γίνει και βέβαια θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αν όλοι στην Ευρώπη συμμορφώνονταν με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Είναι λοιπόν σαφές ότι αν κάνουμε κάποιο λάθος μας διορθώνει το δικαστήριο. Και η ε, παρούσα επιτροπή έχει καταχωρήσει όλες τις πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες εκτός από μία που ήταν να σταματήσει το Brexit, για την οποία όμως δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε καταχωρήσει λοιπόν όλες τις πρωτοβουλίες Κάποιες φορές εν μέρη μια καινοτομία που ε, εισήγαγε η Επιτροπή μας με βάση τις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου. Νομίζω άλλωστε ότι όλοι έχετε επικροτήσει αυτή την ιδέα της μερικής καταχώρησης. Ε, και ο κύριος Γκένος νομίζω αναφέρθηκε στο θέμα του τμήματος που δεν καταχωρίζεται. Δεν είμαι βέβαιος αν αυτό θα πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν ε, αυτό θα γίνεται από τις επιμέρους αρχές, αλλά θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Ο κύριος Σέπφλιν επίσης ρώτησε ποιες ήταν οι τέσσερις πρωτοβουλίες πολιτών ε, και ήταν ε, το δικαίωμα στο νερό, η γλυφοσάτη, ε, το να σταματήσουν τα πειράματα σε ζωντανά ζώα και... Και όσον αφορά τη δημόσια διαβούλευση, 5.000 απαντήσεις λάβαμε, το 96% αυτών ήρθαν από πολίτες και αποτέλεσαν σημαντική συνεισφορά στην πρόταση που υποβάλαμε, ιδιαίτερα όσον αφορά το πόσο πολύπλοκη ήταν η καταχώρηση και η παρακολούθηση των εξελίξεων. Θεωρήσαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να είμαστε πάροχος υπηρεσιών στο θέμα αυτό. Επίσης προτείναμε περίοδο παρακολούθησης πέντε μηνών αντί για 3 μήνες για να υπάρχει περιθώριο για συζήτηση. Διότι και αυτό ήταν μια από τις προτάσεις που λάβαμε και θα είχαμε έτσι τη δυνατότητα να αντιδράσουμε με τρόπο πιο λογικό και επικοδομητικό. Επίσης, Σκοπό είχαμε να ε, παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ε, και να δημιουργήσουμε σχετική πλατφόρμα. Ας μην θεωρούμε όμως ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών είναι η πανάκια για την Ευρώπη. Είναι ένα λιθαράκι στο τείχος, στα θεμέλια που θα πρέπει να χτίσουμε της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Μην παραδιαφημίζουμε λοιπόν κιόλα ε, το ε, εργαλείο αυτό και σα το λέω αυτό ως ε, ένα από του ανθρώπου που έλαβαν την πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει, όχι όμως να νομοθετήσει. Εάν συγκεντρώσουμε τα δεδομένα με βάση την εθνικότητα, νομίζω ότι ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο των διπλών υπογραφών διατηρώντας και μια καλή ισορροπία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δεσμευτικό το μέσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε πολίτες σε, δύο χώρες να... Μάλλον ένας πολίτης να κατοχωριστεί σε δύο χώρες. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη πρόταση για να το αποφύγουμε αυτό. Το να έχουμε δύο έντυπα δηλαδή και νομίζω ότι έτσι είναι πιο σαφή τα πράγματα. Τώρα, πώς υποστηρίζουμε τους διοργανωτές. Θα υπάρχει ένα help desk το οποίο θα είναι χρήσιμο, θα υπάρχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα αλληλεπίδραση, θα υπάρχουν και ε, μεμονωμένα σημεία επαφή ε, στα κράτη-μέλη. Και όλα αυτά, όπω γνωρίζετε, επειδή συνέβη και εδώ στο κτίριο, ε, είναι πράγματα τα οποία πρότειναν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει που συμμετείχαν στι πρωτοβουλίε των πολιτών. Ήταν πράγματα τα οποία επιθυμούσαν και νομίζω ότι είχαμε και θετικέ απαντήσει από αυτού και χαίρομαι που το λέω. Και πάλι λοιπόν, όπως σας είπα, όταν ε, το δικαστήριο ε, σου σε επιπλήττει ε, το αντιλαμβανόμαστε και το δεχόμαστε. Το είχαμε για το Stop TTIP και για το Minority Safe Pack και τώρα προσέχουμε περισσότερο τις αποφάσεις μας παρεπιπτόντων σαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω το είπε ο κύριος Ντουράν αυτό, θέλει να ε, έχει ψήφισμα για τα θέματα αυτά, γιατί όχι, αυτό επαφείται σε εσά. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Αν θέλετε να έχετε ψήφισμα ή συζήτηση, εγώ εδώ είμαι. Ή όποιο θα είναι αρμόδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα. Αλλά αυτό επαφείται σε εσά. Ε, και φυσικά εμείς ε, θα απαντήσουμε θετικά στο σχετικό αίτημα. Όσον αφορά την χρηματοοικονομική υποστήριξη για τους διοργανωτές. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο θέμα διότι ε, η αρχή της εξαρτησίας της πρωτοβουλίας των πολιτών θέλουμε να διατηρηθεί. Αν αρχίσουμε να παρέχουμε χρηματική υποστήριξη μπορεί να υπάρξουν ερωτηματικά ε, για την ε, αρχή της ανεξαρτησίας και φυσικά μπορεί να επιβαρύνει και περισσότερο τους διοργανητές. Θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις για το πώς δαπανήθηκαν τα κονδύλια. Ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και θέλουμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες, όχι να τις περιπλέξουμε. πέραν αυτού, ναι μεν δεν ε, προσφέρουμε χρηματοοικονομική υποστήριξη, αλλά προσφέρουμε σε είδο. Ε, δίνονται συμβουλές, υπηρεσίες μετάφρασης, ε, δωρεάν διαδικτυακό σύστημα συλλογής υπογραφών και νομίζω ότι αυτό θα μειώσει το άφθο για τους οργανωτές. Η διαφάνεια, το ρώτησαν και ο κύριος Βαλέσα και άλλοι, ε, θέλουμε οι διοργανωτές να δίνουν επικαιροποιημένες ε, ε, πληροφορίες για όλες τις πηγές χρηματοδότησης που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ το χρόνο και να υπάρχει απάντηση για την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην δική τους την ιστοσελίδα. Όλα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας των Πολιτών και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε και κάποια μέτρα επιπλέον για να αυξήσουμε τη διαφάνεια ώστε να μην υπάρχουν κατακρίσεις για το θέμα της απαγόρευσης της γλυφοσάτης. Εδώ θα πρέπει να είμαι απόλυτα σαφής. Η απαγόρευση της γλυφοσάτης για να προστατεύσουμε τους πολίτες και το περιβάλλον για τα τοξικά ε, φυτοφάρμακα είναι η τέταρτη πρωτοβουλία των πολιτών που απαιτούσε ένα εκατομμύριο υπογραφέ από τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη. Υπευλήθη επισήμως σε εμά στις 6 Οκτωβρίου και έκτοτε στις 23 Οκτωβρίου συναντηθήκαμε επισήμως με τους διοργανωτές του πρωτοβουλίας για να μας εξηγήσουν πολύ αναλυτικά τα θέματα της πρωτοβουλίας. Στις 20 Νοεμβρίου έγινε δημόσια κρόαση για το θέμα εδώ. Η αναθεώρηση της έγκρισης της γλυφοσάτης βάσει του κανονισμού των φυτοφαρμάκων είχε ήδη προχωρήσει όταν απεστάλει πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 27 Νοεμβρίου γνωρίζετε ότι ε, η αρμόδια επιτροπή κατέληξε σε συμφωνία για ανανέωση για πέντε χρόνια ακόμα. Και έτσι θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, η πρωτοβουλία πολιτών δεν αφορά μόνο τη γλυφοσάτη, αλλά καλύπτει και άλλα θέματα πολιτικής φυτοφαρμάκων και εγκρίσεων φυτοφαρμάκων και τη διαδικασία της έγκρισης αυτών των ουσιών. Αυτή τη στιγμή ε, εκπονείται μία ανακοίνωση για τα συμπεράσματα για αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τι δράση θα αναλυφθεί εάν αναλυφθεί και για ποιο λόγο θα αναλυφθεί ή όχι δράση. Όπως σας είπα, προσέχουμε πάρα πολύ και εξετάζουμε πάρα πολύ δεξιωτικά την αιτιολόγησή μας. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες επ' αυτού, διότι πρέπει να τα εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά σε εσωτερικό επίπεδο επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προθεσμία για να απαντήσουμε είναι 8 Ιανουαρίου, από ό,τι φαντάζομαι θα εγκριθεί η απάντησή μας μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα, ε, τελευταία παρατήρηση, γιατί και εγώ δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να επανέλθω και στα όσα είπε ο κύριος Έπφλιμ, Βαλέσα και άλλοι. Υπάρχει το θέμα δηλαδή το τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία. Και εκεί θα ήθελα να σας καλέσω να μας βοηθήσετε να τη βελτιώσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι και η βασική μας επιθυμία. Ας μην λοιπόν προσπαθούμε να το παρουσιάσουμε ως ένα εργαλείο άμεσης δημοκρατίας που δίνουν στους πολίτες δυνατότητα να επηρεάσουν άμεσα την νομοθεσία. Όχι. Κανείς από τους εισηγητές στο Κοινοβούλιο δεν έκανε κάτι τέτοιο και όλοι είναι ξεκάθαροι για το τι έχουμε εδώ. Βρισκόμαστε ήδη όλοι ε, στην ίδια σελίδα, παρόλο που μπορεί να μην συμφωνούμε σε κάθε μια γραμμή. Και είναι η ευθύνη του να εξηγήσουμε ποιος είναι ο ρόλος, σε ποιο, ποιο στόχο εξυπηρετεί και εμείς εδώ επικυρώσαμε τη συνθήκη. Και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα προκάλεσε ένα εκνευρισμό τα τελευταία πέντε χρόνια, που είναι η περιπλοκότητα της όλης διαδικασίας και το γεγονός ότι δεν γίνεται καθόλου feedback μετά, έχουν να κάνουν με την ε, έλλειψη απόκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βελτιώνουμε και χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω προσπάθειες. Και αν το φτιάξουμε, πιστεύω πως ο κόσμος θα καταλάβει πως παρόλο που πώς θα καταλάβουν πώς. Μπορεί να μην συμφωνούν μαζί μας στην απόφαση που τα λαμβάνουμε κάθε φορά, αλλά αν έχουν feedback από εμάς θα καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχουμε κάνει και το βάρος απόδειξης βέβαια είναι δικό μας. Δεν το κάνουμε πάντα στο παρελθόν, θα το κάνουμε όμως, σας το εξασφαλίζω στο μέλλον και νομίζω ότι αυτή, αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη θητεία θα πάει καλύτερα από τους προηγούμενους με αλλαγές στον κανονισμό και νομίζω πως θα τα πάμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον και παραμένω στη διάθεσή σας και στη διάθεση όλων των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο με τροπολογίες όπου κρυθεί απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ όλες τις επιτροπές που συμμετείχαν σε μια πολύ ε, καλή συζήτηση και θα ήθελα τώρα εγώ να στραφώ προς τα μέλη μου και να σας πω πως θα πρέπει να επιστρέψουμε στην αίθουσα της Επιτροπής που ήμασταν σήμερα το πρωί. Είμαι πεπισμένη πως οι δύο επιτροπές μας θα βοηθήσουν στο να εγκρίνουμε τον νέο κανονισμό πριν το τέλος της τρέχουσας θητείας του Κοινοβουλίου. Ας είμαστε λοιπόν σε επαφή και συνεχίσουμε την καλή δουλειά. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. So. no, no, no. Just in case. Okay. okay, thank you. So, colleague, if you want to take a seat, no, no, it's, it's, it's open. It's open. Καθίστε, συνάδελφοι, είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Κύριε Λαμασούρ, σας παρακαλώ καθίστε. Ευχαριστώ. We can start. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η Ντανούτα Χούπνερ ζητά συγγνώμη, θα έρθει λίγο αργότερα και θα ξεκινήσω εγώ με το εργαστήριο για τις συνέπειες του Brexit στα Ιρλανδικά σύνορα. Ένα πολύ δύσκολο θέμα. Όπως γνωρίζετε έχουμε τέσσερις παρεμβάσεις, μία από δύο διαφορετικούς ανθρώπους, είναι τρεις δηλαδή παρεμβάσει παρεμβάσεις συνολικά, αλλά θα ακούσουμε τέσσερις ομιλητές. Οι δύο που θα ξεκινήσουν είναι ο καθηγητής ε, David Finmore και η ε, καθηγήτρια Katie Hayward. αν κατάλαβα καλά, η κυρία Hayward θα ξεκινήσει και μετά θα λάβει το λόγο ο κύριος Finmore. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το θέμα σήμερα και παρόλο που φτάνουμε στην 20η επέτειο της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής αυτή τη στιγμή δεν τη θεωρούμε ως ένα ιστορικό έγγραφο αλλά ως μια ζωντανή και δυναμική συμφωνία και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως και ο Ντέιβιτ και εγώ ε, διδάσκουμε φοιτητές οι οποίοι έχουν μεγαλώσει ε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία ε, και έχουν ανδρωθεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πρόκειται λοιπόν ε, για ένα έγγραφο από το παρελθόν, αλλά για ένα δυναμικό έγγραφο μέσα σε μια εύθραυστη ειρήνη ε, που ε, βιώνουμε αυτή τη στιγμή στο Μπέλφαστ, Οπότε μπορώ να σας πω ότι επειδή έχει και δύο ονόματα είναι η Συμφωνία του Μπέλφαστ ή η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Και αυτό αποδεικνύει και πόσο εύθραυστη είναι. Από το 98 και μετά που υπεγράφει έχει ενισχυθεί με άλλες συμφωνίες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ε, έχουν υπογράψει τις συμφωνίες αυτές που βασίζονται στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Έχουμε πάρα, πολλά, πάρα πολλές λεπτομέρειες στην έκθεση που καταθέσαμε και στην παρουσίασή μου απλώς θα περιγράψω τους βασικούς λόγους για τους οποίους είναι τόσο σημαντικό το Brexit για τη συμφωνία αυτή. Και μετά ο David θα μιλήσει και για κάποιες από τις λύσεις που ενδεχομένω μπορούν να εφαρμοστούν. Να σας πω καταρχήν πώς περιγράφεται η σύραξη στη συμφωνία. Στο κείμενο το ίδιο βλέπουμε πως ορίζεται ως μία σύραξη μεταξύ δύο παραδόσεων. Δεν λέμε καθολικοί και προτεστάντες, αλλά λέμε ενωτικοί ε, και εθνικιστές, γιατί είναι οι ταυτότητες αυτές και οι πολιτισμοί αυτοί και οι ιστορίες αυτές και οι πολιτικές προσδοκίες, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ αυτών των δύο παραδόσεων και εκπροσωπούνται και στηρίζονται από το κράτος της Ιρλανδίας και το κράτος της Βρετανίας. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι πολιτικές προσδοκίες και ταυτότητες να θεωρούνται εξίσου νόμιμες. Και η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας είναι ουσιαστική και πάνω σε αυτό βασίζεται η επιτυχία της ίδιας συμφωνίας. Έχουμε κάποιες βασικές αρχές, οπότε θα αναφερθώ σε κάποιες από αυτές. Καταρχήν, η αυτοδιάθεση για τους λαούς του, της νήσου της Ιρλανδίας. Και εδώ θα ήθελα να συμπιστήσω την προσοχή στο ότι η ειρήνη στη Βόρεια Ιρλανδία δεν αποτελεί εγχώριο θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου και η Ιρλανδία, ε, το κράτος, η δημοκρατία της Ιρλανδίας και ο Ιρλανδικός λαός εμπλέκονται. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε τη συνένεση της πλειοψηφίας, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή στη συνταγματική τάξη της Βορείου Ιρλανδίας θα πρέπει να εγκριθεί μέσω ε, πλειοψηφίας στην Βόρειο Ιρλανδία, όπως επίσης και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Δηλαδή, τις αλυτρωτικές ε, τάσεις που είχε η, το, η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ε, από το παρελθόν τις έχει αποσύρει. Ένα ακόμα καλό στοιχείο ότι βασίζεται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζεται πολύ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και βασίζεται στο ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη Βόρεια Ιρλανδία ως ένα μεμονωμένο θέμα. Έχουμε τα τρία στελέχη αυτής της συμφωνίας που είναι ο Βορράς και ο Νότος στο νησί της Ιρλανδίας και Ανατολή Δύση γιατί βέβαια υπάρχει η Βρετανία και η Ιρλανδία. Είναι ε, λοιπόν αλληλεξαρτούμενα και οποιαδήποτε λύση για το μέλλον θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτή την αρχή. Θέλω να περιγράψω στα γρήγορα τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμφωνία. Όπως λέμε και εμεί στην έκθεση, οι αναφορές που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κείμενο της Συμφωνία, είναι ε, άσχετες με το θέμα μας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, σκεφτήκαμε τη συμφωνία αυτή. Αποτελεί δηλαδή ένα μοντέλο και ένα πλαίσιο για την επιτυχία της ίδιας συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι παρόλο που δεν έχει κάποιον υποχρεωτικό ρόλο, δεν έχει ούτε το καρότο ούτε το μαστίγιο, παρόλα αυτά έχει ένα πολύ ορατό και σημαντικό ρόλο που είναι αυτού που διευκολύνει. Και θα ήταν αδιανόητο να υπογράψουμε τη συμφωνία αυτή χωρίς το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αξιοσημείωτο πως την δήλωση στήριξης αυτής της συμφωνίας, όπως επίσης και στην δήλωση στήριξης της Αγγλο-Ιρλανδικής Συμφωνίας του 1995, η Ιρλανδία και η Βρετανία αναφέρονται στις σχέσεις τους ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πόσο κομβική σημασία είναι η σχέση αυτή. Στη διαδικασία της διασυνοριακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, ε, να σας πω πως το σημείο αυτό ήταν σημαντικό για τις στενές και παραγωγικές σχέσεις που έχει ολόκληρο το νησί μεταξύ του αλλά και η Ιρλανδία με τη Βρετανία και έχει βασιστεί σε αμοιβαία συμφέροντα, αμοιβαία πλεονεκτήματα και είναι αποπολιτικοποιημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο το οποίο προσέφερε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πως αποτελεί ως κίνητρο για την για ολόκληρη την οικονομία του νησιού της Ιρλανδίας με την προσπάθεια σύγκλησης μεταξύ βορρά και νότου. Τέλος, για να εντοπίσω κάποιες από τις βασικές προκλήσεις που ε, δημιουργεί το Brexit, καταρχήν να σας πω πως ήδη βλέπουμε πως το Brexit δημιουργεί κάποια αστάθεια στην διαδικασία ειρήνευσης και πιο συγκεκριμένα δημιουργεί πόλωση. Και αυτό κυρίως επειδή οι επιλογές που δίδονται Δηλαδή θα πρέπει είτε να μετακινηθεί η Βόρεια Ιρλανδία ε, εγκύτερα στην ε, Βρετανία είτε στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας δημιουργεί μια ε, διπλή, δική επιλογή την οποία είχαμε ξεπεράσει μέσω της συμφωνίας και η οποία αποτελεί ανάθεμα για την ειρήνευση στη Βόρεια Ιρλανδία. Δηλαδή το να θέτουμε αυτή την εναλλακτική ή e ή e ε, απομακρύνεται από τις βασικές αρχές επί τις οποίες υπογράφει και η συμφωνία. Δεύτερη ε, βασική πρόκληση είναι η ίδια συνοριακή ε, συνεργασία και πώς αυτή έχει επαναπολιτικοποιηθεί και είναι δύσκολο να δούμε πώς θα εξομαλυνθεί ή θα αποτελέσει πλέον κομμάτι της καθημερινής δραστηριότητας. Και αυτό δημιουργεί πολλές προκλήσεις για την επιτυχία και τη σταθερότητα της συμφωνίας. Και τέλος, η συμφωνία βασίζεται στην ισότητα μεταξύ Ιρλανδών και Βρετανών πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία και την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Οποιαδήποτε πρόκληση προς αυτή την αρχή δημιουργεί κίνδυνο για την ίδια συμφωνία και για την διαδικασία ειρήνευσης. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Okay. Um, it's to me to offer some of the σας παρουσιάσω κάποιες από τις προτάσεις ε, στην μελέτη μας σχετικά με το πώς μπορεί να ε, συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και λέω να συνεχίσει να ισχύει, διότι υπάρχει η άλλη πτυχή εξίσου ε, σημαντική. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το πλαίσιο για συνέχιση της ισχύω της συμφωνίας. Και θέλω να μιλήσω και σε ε, γενικότερο επίπεδο και όσον αφορά τις ε, διασυνοριακές πτυχές. Για τη διατήρηση της ε, συμφωνίας υπάρχει σαφής προόδος στις δεσμεύσεις και του Ηνωμένου Βασιλείου και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζεται η συμβολή της συμφωνίας στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Επίσης, υπάρχει η επιθυμία, η βούληση τουλάχιστον ε, να ακολουθηθούν ε, καινοτόμες ε, λύσεις. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με κάποιες από τις προκλήσεις που ανέφερε η συνάδελφος. Όσον αφορά την ίδια την συμφωνία, νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι τομείς όπου θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορεί να γίνει ώστε τις δεσμεύσεις αυτές να τις κάνουμε πράξη μπορεί όχι μόνο να αναγνωρίσει, αλλά προστατεύσει κανείς τα δικαιώματα ε, Ιρλανδών πολιτών ε, στην Βόρεια Ιρλανδία. Μπορεί να παίξει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιο ρόλο. Πώς θα διατηρήσουμε ε, την εκπροσώπηση των Ιρλανδών της Βόρειας Ιρλανδίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούν, θα ίσως να ψηφίζουν ε, σύμφωνα με τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Και επίσης στο έγγραφό μας λέμε ότι θέλουμε να εξετάσουμε τον ρόλο κλειδί των θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο της, διαδικα... της συμφωνίας διότι το μέλλον της συμφωνίας αυτής ε, έγκυται και στην, ε, στο να εκμεταλλευτούμε ε, πλήρως την ίδια την συμφωνία. Ωστόσο, η βασική μας πρόκληση είναι να διατηρήσουμε το πλαίσιο για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην παροχή των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της συμφωνίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου έχουμε καταρχάς ε, την ελαχιστοποίηση ε, των ε, αναταράξεων όσον αφορά την οικονομική ζωή στη Βόρεια Ιρλανδία και εδώ έχει να παίξει σημαντικό ρόλο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεύτερον, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε όσο γίνεται προσπελάσιμα σύνορα, όσο σήμερα δηλαδή. Τρίτον, θα πρέπει να διατηρηθεί το νομικό και οικονομικό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να διατηρήσουμε τις ευκαιρίες που παρέχονται σήμερα για ε, θεσμική διασυνοριακή συνεργασία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς προτείνουμε διάφορες ιδέες στο έγγραφό μας που βασίζονται σε ιδέες άλλων ε, γύρω από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Βέβαια, αν είχαμε συμπεριλάβει τα πάντα, το έγγραφό μα θα είχε το διπλάσιο μέγεθος. Σημαντικό πάντως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει τέτοια σχέση με, το, με την Ευρωπαϊκή Ένωση που να προσωμιάζει όσο γίνεται περισσότερο στο status quo. Κυρίως ε, να παραμείνει μέρος ε, της Τελωνιακής Ένωσης ε, και της Εσωτερικής Αγοράς. Εναλλακτικά προτάθηκε η Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να έχει ειδικό καθεστώς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εμείς αναγνωρίζουμε στο εγγραφό μας ότι δεν υπάρχει πολύ πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποιο είδους διακριτικής μεταχείρισης της Βόρειας Ιρλανδίας στο πλαίσιο του Brexit και θα πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχουν εάν υπάρχει δυνατότητα να παραμείνει η Βόρεια Ιρλανδία ε, στην εσωτερική αγορά μέσω συμμετοχή, για παράδειγμα, στον ε, ΕΟΧ. Αυτό όμω δεν θα αποτελέσει πανάκια για τι προκλήσει ε, του Brexit στη Βόρεια Ιρλανδία διότι θα υπάρχει ακόμα το θέμα των συνοριακών ελέγχων κατά την διακίνηση αγαθών. Το θέμα λοιπόν είναι, μπορεί να παραμείνει εντό Θελωνιακή Ένωση η Βόρεια Ιρλανδία ή να έχει κάποια ειδική θελωνιακή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμω δεν λύνει το θέμα του εμπορίου γεωργικών προϊόντων που είναι τόσο σημαντικό για διάφορε περιοχέ τη Βόρεια Ιρλανδία και ιδιαίτερα τι μαθοριακέ περιοχέ. Θα μπορούσαν έτσι λοιπόν να υπάρξουν ε, οι ρυθμίσεις ε, ώστε η Βόρεια Ιρλανδία να υποφελείται πλήρως από το εμπόριο, τουλάχιστον στην ίσο της Ιρλανδίας, αν όχι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικά πολιτικά θέματα και προκλήσεις ε, που συνδέονται με τις λύσεις αυτές. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο ανυπέρβλητο νομικό εμπόδιο για να το πετύχουμε αυτό. Είναι καθαρά θέμα πολιτικών προτιμήσεων και πολιτικής βούλησης. Εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία από αυτές τις λύσεις, ε, τότε τι θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε. Νομίζω ότι σημαντικό εδώ πέρα είναι να επικεντρωθούμε σε δύο πράγματα. Καταρχάς, να διατηρήσουμε όσο γίνεται πιο προσπελάσιμα σύνορα. Αυτό είναι ζωτική σημασία ε, για την οικονομία, αλλά και για την ε, συνέχιση της εφαρμογής ε, της ε, συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και της ειρηνευτικής διαδικασίας. Εδώ λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όσον αφορά την διακίνηση αγαθών και θα ακούσουμε από τον κύριο Λάρς Κάρλσον πώς μπορούν από τεχνικής άποψης να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Αλλά όσον αφορά την Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να το να επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε τεχνικές λύσεις δεν είναι ιδανικό. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ειδική φύση, γεωγραφική και πολιτική των συνόρων στη Βόρεια Ιρλανδία και τη σημασία του διασυνοριακού εμπορίου για την οικονομία. Πέρα από το εμπόριο όμως, νομίζω ότι σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε τον ρόλο που έχουν παίξει μέχρι τώρα τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την ευημερία στη Βόρεια Ιρλανδία, για την ε, υποστήριξη αγορών που καλύπτουν το σύνολο του νησιού, καθώς και για τη συνεργασία βορρά και νότου στο νησί. Θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε αυτά τα βασικά στοιχεία της ειρηνευτικής διαδικασίας και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους πρόσβαση ε, της Βόρειας Ιρλανδίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ε, είτε μιλάμε για το, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε για το Ίντερνετ, είτε για άλλα προγράμματα. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος διασυνοριακά προγράμματα για το σύνολο του νησιού να μπορούν να ε, συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά. Ή να θεωρηθεί το βόρειο τμήμα του νησιού επίση Ιρλανδικό ε, για του σκοπού των προγραμμάτων αυτών. Αυτέ είναι ιδέε που έχουμε αναπτύξει στο εγγραφό μα ε, και θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθούν καινοτόμε λύσει για να αντιμετωπιστούν κάποιε από τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Βόρεια Ιρλανδία ε, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερις παρατηρήσεις ε, ως συμπεράσματα. Καταρχάς θα πρέπει να διατηρήσουμε το πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεύτερον, θα πρέπει να φροντίσουμε τα σύνορα να παραμείνουν όσο γίνεται πιο προσπελάσιμα. Τρίτον, θα πρέπει η Βόρεια Ιρλανδία να θεωρηθεί κόμβος επαφών ε, ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ε, εδαφικές ε, διαφορές και να χρησιμοποιήσουμε καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις για να αποφύγουμε όσο γίνεται αλλαγές στο status quo και να έχουμε έτσι επιτυχία εφαρμογή στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίνιμορ και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στον ε, καθηγητή Λάρς Κάρστελ. Εσείς είστε ο άνθρωπος που ασχολείται με τα σύνορα και τα τελωνία. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρακτικές λύσεις και αυτά θα μας δώσετε στην παρέμβασή σας. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Ε, είναι τιμή, προνόμιο και χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να σας απευθύνω το λόγο για τα ευφυή e e σύνορα εκδοχή 2. Και πράγματι εγώ είμαι άνθρωπος των τελωνίων, ασχολούμαι με την τελωνιακή πολιτική και την πολιτική συνόρων για πάνω από 30 χρόνια και ασχολούμαι σε πάνω από 180 χώρες και έχω δει πάνω από χίλια σύνορα και πραγματικά ε, θα μιλήσω για θέματα σύνορων και των δελωνίων στα επόμενα λεπτά. Θα ξεκινήσω όμως με κάτι άλλο. Στις 14 ε, Απριλίου 1970 ε, είχαμε τη διάσημη φράση «Χιούστον έχουμε πρόβλημα» και τώρα χρησιμοποιείται ε, ως ε, ε, μήνυμα όταν μας περιμένουν μεγάλα προβλήματα. Και επομένως και εγώ θα πω Βρυξέλλες, Λονδίνο έχουμε πρόβλημα ο κυβερνήτης του Απόλλω 13 τελικά κατάφερε να προσγειώσει ε, το Απόλλω 13 και χρησιμοποίησε τις δεξιότητες, την εμπειρία του και τις τεχνικές του γνώσεις για να μπορέσει να προσγειώσει το αεροσκάφος και να ε, φέρει το πλήρωμα πίσω ε, και το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς ε, στα θέματα της διαχείρισης ε, των συνόρων διότι υπάρχουν και καλά και άσχημα νέα. Πάντα ξεκινώ με τα άσχημα νέα διότι θέλουμε στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε με τα καλά νέα. Όταν κάποιος φεύγει από κάπου σημαίνει ότι φεύγει και από την τελωνιακή επικράτεια. Και αυτό που γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ε, τα τελευταία 30 χρόνια είναι ότι όταν υπάρχει αποχώρηση ε, σημαίνει ότι ε, έχουμε Πανεγκατάσταση συνόρων και αυτό φυσικά θα γίνει. Το θέμα που μας αποσχολεί είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα ωφέλη της διαχείρισης των συνόρων αυτών με έναν ευφυή, σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο. Τα καλά νέα είναι ότι αν εξετάσουμε τα σύνορα της Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας και οι συνάδελφοι στο πάνελ τα παρουσίασαν και αυτοί στην εκθεσή τους, είναι ένα ε, σύνορο ζωτικής σημασίας. Μπορεί να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ε, ε, κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών και είναι ουσιαστική αυτή η κυκλοφορία και πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση που θα μπορέσει ε, να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Τα καλά νέα είναι ότι ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε αυτά από πρακτική πλευρά, διότι πριν από 50 χρόνια δεν ξέραμε τι ήταν η παγκοσμιοποίηση. Τώρα γνωρίζουμε την παγκοσμιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση είναι αυτή η οποία οδηγεί την εναρμόνιση. Σήμερα υπάρχουν διεθνή πρότυπα στον τομέα των τελωνίων και των συνόρων, τα οποία παρέχουν μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν λειτουργικά αυτά τα σύνορα ε, και να είναι όσο το δυνατόν πιο ε, αόρατα, αλλά φυσικά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, ε, διότι πρέπει να γίνει η διαχείριση των συνόρων και η διαχείριση των συνόρων δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο για τους λόγους που διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, ένα από τα προφανή που σκεφτόμαστε πάντα όλοι είναι ε, να συλλέγονται δασμοί και φόροι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους γίνεται η διαχείριση των συνόρων, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Υπάρχουν θέματα ασφαλείας, θέματα προστασίας, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αγαθά με διαφορετικό καθεστώς και πώς κινούνται ε, από το ένα σύνορο στο άλλο και γιατί πρέπει να γίνεται διαχείριση των σύνορων ανεξάρτητα από θέματα ε, δασμών και φόρων που επιβάλλονται. Όταν λέμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τον τάδε δασμό ή να υπάρξει η τάδε εμπορική συμφωνία, δεν σημαίνει ότι ούτω ή άλλω δεν πρέπει να γίνει διαχείριση συνόρων. άλλως δεν πρεπει να γίνει με διαφορετικούς τρόπους και αυτό είναι που έχει σημασία τελικά. Αυτό το οποίο εξετάζουμε και αυτό που εξετάζω και εγώ στην έκθεσή μου είναι ποιες είναι τα, ποια είναι τα παραδείγματα που έχουμε από βέλτες πρακτικές. Υπάρχουν διεθνή πρότυπα, επομένως θα υπάρχουν και παραδείγματα από βέλτες πρακτικές και όντως υπάρχουν. Εξετάζουμε λοιπόν διάφορα καλά παραδείγματα σε αυτή την έκθεση και θέλουμε να προωθήσουμε. Ε, δεν ε, χρειάζεται να σας δώσω λεπτομέρειες, μπορείτε να τα διαβάσετε, υπάρχουν στην έκθεση. Ένα καλό παράδειγμα είναι τα συνορα Σουηδία Σουηδίας-Νορβηγίας που διαχειρίζονται όλα τα, τα θέματα τα οποία σας αναφέρω με πολύ ομαλό, ε, γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν χρησιμοποιήσει πολλά από τα συστατικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διαχείριση συνόρων και ε, επίσης αυτό που ισχύει είναι ότι ε, αυτό είναι και εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Νορβηγία σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό που ε, λέω είναι ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις στα συγκεκριμένα αυτά σύνορα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένως ε, στα σύνορα Ιρλανδίας-Βόρειας Ιρλανδίας. Και να πω ήδη εκ των προτέρων ότι παρά το γεγονός ότι κάποιοι από τους συναδέλφους, ο καθηγητής Φίνεμορ και Χέιουαρντ αλλά και ο καθηγητής Δομπελάνη εξετάζουν αυτό το συγκεκριμένο θέμα περισσότερο από πλευράς πολιτικής, από πολιτική σκοπιά ε, και μπορεί να υπάρξει ίσως και κάποια μακροοικονομική αντιμετώπιση. Εγώ θα ήθελα επίσης ε, να θίξω και το θέμα ε, της τεχνικής πτυχής, διότι υπάρχει και τεχνική πτυχή. Κάποιοι συνάδελφοι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι και δεν πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να τα καταφέρουμε. Εγώ είμαι πολύ πιο αισιόδοξο. και αυτό είναι θέμα συζήτησης τα συνορα Σουηδία Νορβηγία έχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε πλαισιο βόρεια Βόρειας Ιρλανδίας-Ιρλανδίας. Το αυτό ισχύει και για τα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και καλύπτουν πολλά από τα διεθνή πρότυπα και χρησιμοποιούν τα μοντέλα τα οποία συζητούμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Τρίτο παράδειγμα το οποίο εξετάσαμε είναι ενδιαφέρον παράδειγμα και θα μπορούσε να ρωτήσει κανεί γιατί το εξετάσουμε. Είναι τα σύνορα Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία. Ε, δεν έχουν χερσαία σύνορα, αλλά ε, διαθέτουν κάποια από τα στοιχεία των διεθνών προτύπων τα οποία εφαρμόζονται και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε μια νέα εκδοχή αυτών των συγκεκριμένων σύνορων το οποίο μας φέρνει στα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται. Ε, θα, ε, θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, παρόλο που θα μπορούσα, ε, θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ μέχρι αύριο, αλλά εγώ δεν έχω τόσο χρόνο. Υπάρχουν κάποια διεθνή πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν εφαρμοστεί παντού πλήρως. Και ένα από τους λόγους για τους οποίους σήμερα υπάρχει ο ΠΟΕ και η Συμφωνία Διευκόλυνση Εμπορίου του ΠΟΕ είναι για να εφαρμοστούν πλήρως αυτά τα πρότυπα στην οικονομία μας. Πρόκειται για μια διαδικασία δηλαδή η οποία να είδε εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η χρήση λοιπόν αυτών των συστημάτων και μάλιστα με αναβαθμισμένο τρόπο, καλύτερα και με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Και εδώ ερχόμαστε στα έξυπνα σύνορα. Πρόκειται για μία έννοια η οποία εμφανίστηκε πριν από 15 χρόνια περίπου στην ε, Βόρεια Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη και έχει ε, κάποια διακριτικά χαρακτηριστικά. Καταρχάς ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα διεθνή πρότυπα τα οποία υπάρχουν ήδη. Το δεύτερο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το συγκεκριμένο είναι να χρησιμοποιηθεί συντονισμό, που σημαίνει να τον δούμε από δύο σκοπιές. Ε, καταρχάς συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών από τη μια πλευρά των συνόρων και επίση συντονισμό και των δύο πλευρών ε, που βρίσκονται κατά έρωθεν των συνόρων. Δηλαδή να μην ε, διπλασιάζονται όλα από τι απαιτήσει ε, για πληροφορίε ή του ελέγχου όταν πρέπει να υπάρχουν έλεγχη. Το τρίτο στοιχείο είναι η του ελεγχου οταν κινδύνου. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στη διαχείριση κινδύνου η Μπορούμε πάντα να βελτιωθούμε, αλλά είναι τμήμα τη έννοια των έξυπνων συνόρων. Να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα βάσει αξιολόγηση κινδύνων. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα έξυπνα σύνορα ε, μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξουμε τα απαραίτητα πράγματα που πρέπει να ισχύουν στα σύνορα, ανεξάρτητα αν θέλουμε να είναι προσπελάσιμα ή μη και θα, πρέπει να γίνουν πριν ή μετά τα σύνορα. Αυτά τα συγκεκριμένα καθεστώτα συμμόρφωσης αναπτύχθηκαν πολύ την τελευταία δεκαετία και πολλά τέτοια διεθνή πρότυπα εφαρμόζονται σε πολλές χώρες και θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν, να απλουστευτούν ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ άλλα συγκεκριμένα ε, στοιχεία. Αυτό το οποίο προτείνω λοιπόν και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι να δούμε και την τεχνική σκοπιά, να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε ε, την ε, δεύτερη εκδοχή των έξυπνων σύνορων. Αντλώντας εμπειρία από τα διεθνή πρότυπα, από τα επιχειρησιακά πρότυπα τα οποία είναι διαθέσιμα ήδη στον κόσμο, να τα βαθμίσουμε, να τα εντάξουμε περισσότερο, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία που είναι απαραίτητη και διαθέσιμη τη σήμερα ημέρα και επίσης να προσπαθήσουμε να τα στήσουμε χρησιμοποιώντα μια σειρά από πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ότι λειτουργούν. Για παράδειγμα, στα σύνορα Σουηδία-Νορβηγία. Για παράδειγμα, τη χρήση μια τεχνική συμφωνία μεταξύ τελωνιακών διοικήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, πληρο... ε, δεδομένων κλπ. Πρέπει να υπάρχουν διάφορε συμφωνίε για το πώ θα συνεργαζόμαστε. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθούν όλα αυτά. Το έχουμε δει αυτό στην πράξη. Αυτά είναι στοιχεία των έξυπνων συνόρων. Δεν θα σας τα αναφέρω όλα γιατί περιλαμβάνονται στην έκθεση, αλλά υπάρχουν. Είναι επιχειρησιακά, λειτουργούν ε, σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Στην πραγματικότητα λοιπόν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά και ε, στα σύνορα Ιρλανδίας-Βόρειας Ιρλανδίας. Και αυτό διότι γνωρίζουμε ότι έχουν αποτέλεσμα αλλά πρέπει να εφαρμοστούν με διαφορετικό τρόπο στα συγκεκριμένα αυτά σύνορα. Ε, κάποιοι μπορεί να πούνε ότι πρέπει να υπάρχει πολλή τεχνολογία ε, και αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολο και δαπανηρό και πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια τεχνολογία. Από τα παραδείγματα όμως που είδαμε στις άλλες μελέτες που έγιναν στην έκθεση μπορούμε να δούμε σαφέστατα ότι υπάρχουν παραδείγματα, για παράδειγμα ε, το παράδειγμα του Gateway το οποίο δοκιμάστηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας, ο πράσινος διάδρομος που χρησιμοποιήθηκε μεταξύ Νορβηγίας και Ανατολικών χωρών και πολλά άλλα παραδείγματα στα οποία υπάρχει ήδη υποδομή η οποία χρησιμοποιείται και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, όπως για παράδειγμα ε, μικροτεχνολογία, διάφορες μορφές κινητής τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες επιλογές από πλευράς τεχνολογίας, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και υπάρχουσες υποδομές για να λειτουργήσουν όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να κατασκευάσουμε παραδοσιακά σύνορα από το μηδέν. Γιατί έτσι λειτουργεί. Αν συμφωνείτε ότι όντω υπάρχουν σύνορα και πρέπει να υπάρχουν τα σύνορα, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τον ίδιο τρόπο που γίνεται παραδοσιακή διαχείριση από τελωνιακέ και άλλε αρχέ. Το συμπέρασμά μου λοιπόν κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι είναι καταρχάς ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι θα υπάρχει σύνορο με τον ένα με τον άλλο τρόπο και πρέπει κάπως να το διαχειριστούμε. Και είναι κοινή ευθύνη να διαχειριστούμε αυτά τα σύνορα, πρέπει να τα διαχειριστούμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνονται. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι να γίνουν αυτά και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο θα είναι ε, στην έννοια των έξυπνων συνόρων που δεν είναι και πυρηνική επιστήμη παρά το γεγονός ότι σας έδωσα το παράδειγμα του Apollo 13 προηγουμένως αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ε, υπάρχουσα γνώση, την υπάρχουσα διεθνή εμπειρία και ε, πάλι τα επιχειρησιακά μοντέλα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Μπορούμε λοιπόν να τα καταφέρουμε, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα υπάρχει δυνατότητα να είναι ομαλή η διαδικασία των συνόρων και να μην είναι ιδιαίτερα επαχθής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνίων, ο ΠΟΕ, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συστήσει όλα αυτά τα μοντέλα. Εμείς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αν θέλουμε και αυτά τα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνίων. Λέει ότι τα σύνορα διαιρούν, τα τελωνία ενώνουν και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε σύνορα με τρόπο που δεν θα ε, δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στα σύνορα ενώ ταυτόχρονα θα γνωρίζουμε και τι περνάει από τα σύνορα για διαφορετικούς λόγους, για να μπορούμε όχι μόνο να τα διαχειριστούμε αυτά τα ώρα τα σύνορα, αλλά να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συμφωνίες που ε, έχουν ε, υποχρέωση να έχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο για να είναι ασφαλές το εμπόριο, να λειτουργεί το εμπόριο και να είναι πιο ασφαλής κόσμος ο κόσμος μας. Ε, και αν μπορούμε να έχουμε μια τεχνική λύση και ένα τεχνικό μοντέλο από κοινού, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα που είναι πολύ πιο ακαθόδη και τελείω διαφορετική φύσεως και είναι διαφορετικό ο τρόπο αντιμετώπισή του με πιο εύκολο τρόπο. Ε, προτείνω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας και να ε, ε προσπαθήσουμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά το συντομότερο. Θα ε, ε, τελειώσω με τον Στίβ Μαριούτσι, τον προπονητή ποδοσφαίρου που είπε πότε θα το κάνουμε, δεν φοράω ρολόι γιατί πάντα Τώρα πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και για την αισιοδοξία σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον καθηγητή κύριο Τεμπελάν που θα μιλήσει για νομικές και οικονομικές πτυχές αυτής της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Οι οικονομίες των δύο τμήματων της Ιρλανδίας είναι πολύ ε, εξαρτώμενος η μία από την άλλη και αυτό υπάρχει, υπάρχει περίπτωση ε, να διαταραχθεί από το Brexit. Η οικονομία της Βόρειας τη Βόρεια Ιρλανδία θα υποφέρει περισσότερο από τον Brexit από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Οπότε η μελλοντική σχέση μεταξύ Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική και για τα δύο κομμάτια τη Ιρλανδίας. Και για τον λόγο αυτό η Ιρλανδική κυβέρνηση δηλώνει πω το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνει στην ενιαία αγορά. Το... Η μελλοντική ευημερία της Βορείου Ιρλανδίας εξαρτάται όχι μόνο και όχι κυρίως από το εμπόριο και τις διευθετήσεις σχετικές για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε τόσο πολύ από το κατά πόσο κάποιο ειδικό καθεστώς, κάποιο είδους θα προβλεφθεί για τη Βόρειο Ιρλανδία. Το μέλλον της Βορείου Ιρλανδίας θα εξαρτηθεί, και μιλώ για το οικονομικό μέλλον, θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα γίνει με την ε, Βρετανική πολιτική σε θέματα γεωργίας στο μέλλον και πιο συγκεκριμένα στις διμερείς συμφωνίες που θα συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο και το κατά πόσο στις συμφωνίες αυτές θα επιτραπούν εισαγωγές φθηνές γεωργικών προϊόντων ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο από άλλες χώρες, τρίτες χώρες από ολόκληρο τον κόσμο. Η άλλη μεγάλη επιρροή για τη μελλοντική ευημερία της Βορείου Ιρλανδίας είναι οποιασδήποτε αποφάσεις ληφθούν στο Λονδίνο μέσα στα επόμενα χρόνια για το κατά πόσο θα έχουμε φυσικές μεταφορές από την Υπουργείο Οικονομικών ε, στο Λονδίνο προς την ε, περιφέρεια της Βορείου Ιρλανδίας. Θα διαπιστώσετε πως από τα πέντε αυτά στοιχεία επιρροής, μόνο δύο ουσιαστικά επηρεάζονται από την άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο θέμα. Και ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας προκαλούν όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα βελτιωθεί, και όλα μοιάζουν ε, να τείνουν να χειροτερεύσουν σε κάποιο βαθμό, μεγαλύτερο ή μικρότερο, αυτό σημαίνει ότι η Βόρεια Ιρλανδία είναι πάρα πολύ ε, ευάλωτη και υπάρχουν και κάποια τμήματα της Δημοκρατίας της που βασίζονται οικονομικά στο εμπόριο με το βόρειο κομμάτι, επίσης κινδυνεύουν και γι' αυτό ανησυχεί τόσο πολύ ο κόσμος. Έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση για τη φύση των συνόρων που θα χρειαζόντουσαν εάν ε, επρόκειτο να συμβούν ε, διάφορα. Το βασικό που πρέπει να σκέφτεστε, γιατί νομίζω ότι δεν έχει τονιστεί αρκετά, είναι πως το πρόβλημα του κατά πόσο ένα σύνορο είναι ορατό ή όχι είναι πολιτικής φύσης. Δεν είναι οικονομικής φύσης. Η ανάγκη σύνορων προκύπτει από τις οικονομικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των οντοτήτων που είναι από τη μία και από την άλλη πλευρά των σύνορων. Οπότε, όταν μιλάτε για ορατά σύνορα, δεν σκέφτεστε για οικονομικά θέματα, αλλά για πολιτικά. Και μία από τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των συνόρων που συζητάμε σήμερα και των συνόρων μεταξύ Σουηδίας και Νορβηγίας είναι πως στην Ιρλανδία δυστυχώς υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και από τις δύο πλευρές των συνόρων ή τουλάχιστον εκεί που θα επρόκειτο να τοποθετηθούν τα σύνορα και κάποιοι από τους λαθρεμπόρους ήταν και ίσως ξαναγίνουν ε, ε, είχαν εμπλακεί και ίσως ξαναεμπλακούν σε παραστρατιωτικές δραστηριότητες. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για οικονομικά θέματα, αλλά μιλάμε και για πολιτικής φύσης θέματα. Και δεν υπάρχει κανένα σύνορο αόρατο ή ορατό, υψηλής τεχνολογίας ή απλό, μπορεί να λύσει τα οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν από μία μη ικανοποιητική οικονομική καθάριση μεταξύ και διευθέτηση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχέση αυτή εξαρτάται από τις διαπραγματεύσει και από τις μελλοντικέ πολιτικές που θα χαράξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν εξαρτάται καθόλου από το κατά πόσο θα υπάρχει ε, φυσικό ή μεταφυσικό σύνορο. Και θα ήθελα να σας τονίσω πως το εμπόριο μεταξύ του, της Βρετανίας ε, και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, του νησιού της Βρετανίας, είναι πολύ πιο σημαντικό σε οικονομικά μεγέθη από αυτό μεταξύ της ε, Βορείου Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Τα ορατά σύνορα, ε, σύνορα με υποδομές, με ελέγχους, με προσωπικό, με κάποιο είδους εξοπλισμό θα χρειαστεί παρόλο που μπορεί σε πολιτικό επίπεδο να μην θέλουμε κάτι τέτοιο, εάν δεν συνάψουν καμία συμφωνία το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, εάν και αυτό που θεωρώ πως είναι το πιο πιθανό για λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, το Ηνωμένο Βασίλειο για τα γεωργικά προϊόντα εγκρίνει μια πολιτική ε, ευθυνών τροφίμων όταν συνάψει συμφωνίε με χώρες, τρίτες χώρες από τον υπόλοιπο κόσμο και επίσης ορατά σύνορα χρειάζονται αν για οποιοδήποτε λόγο το Ηνωμένο Βασίλειο εγκρίνει ε, κανόνες περί φυτοπροστασίας, φυτοϊγιεινής ε, προστασίας ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης από αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα. Το ίδιο ισχύει και αν είναι ε, χαμηλότερο επίπεδο προστασίας για φαρμακευτικά προϊόντα κτλ. Ε, επίσης χρειάζονται φυσικά σύνορα εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρήσει πως είναι ελεύθερο μετά από τις διευθετήσεις που θα κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδοτεί με ελεύθερο και μη ελεγχόμενο τρόπο τις δικές του βιομηχανίες και κλάδους. Μια και φοβάμαι πως όλες οι επιρροές αυτές ενδεχομένως θα γίνουν πραγματικότητα μάλλον δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε τα φυσικά σύνορα εκτός αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα δεχτεί, τουλάχιστον θα δεχτεί να σκεφτεί τουλάχιστον για να λυθεί το θέμα της Βορείου Ιρλανδίας να κάνει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, κα... συναλλαγών κάποιου τύπου όχι ΕΟΧ αλλά κάτι πολύ παρόμοιο μια ελεύθερη ζώνη συναλλαγών μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έδινε τη δυνατότητα στη Βόρεια Ιρλανδία να έχει τα προτερήματα ε, που προσφέρουν και οι δύο δυνατότητες και το ελεύθερο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελεύθερο εμπόριο με το υπόλοιπο του Ηνωμένου Βασιλείου. Βεβαίω εκεί θα υπήρχαν κάποιε απαιτήσει για οποιαδήποτε τέτοιου είδου διευθέτηση, αλλά αν σε πολιτικό επίπεδο μπορούσαν να γίνουν αποδεκτέ, τότε νομίζω ότι δεν θα ήταν δύσκολο από οικονομική άποψη να ε, εγκαθιδρυθούν. Και γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, οι συνάδελφοί μου στο Πανεπιστήμιο Greens προτείνουν αυτό ακριβώς μια λύση ε, ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για τη Βόρεια Ιρλανδία συγκεκριμένα ακόμα και αν το Ηνωμένο Βασίλειο ε, δεν το δεχτεί κάτι που είναι παρόμοιο δηλαδή με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους ομιλητές μας και ιδιαίτερα στους συναδέρφους από το Πανεπιστήμιο Queen's. Ο Δόκτωρ Φένιμορ είναι ένας από τους καθηγητές της κόρης μου και η συμβουλή της προς εμένα σήμερα ήταν «Μαμά, σκέψου προσεκτικά πριν μιλήσεις». Αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, καταρχάς, ε, εισαγωγικά να πω ότι βρίσκομαι εδώ ως ε, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος των Ενωτικών και το λέω αυτό διότι αναφέρεται το κόμμα αυτό στις εκθέσεις. Θα ήθελα να καταστήσω απόλυτα σαφές ότι κανείς στη Βόρεια Ιρλανδία δεν θέλει να επιστρέψει στη βία του παρελθόντος. Κανείς δεν θέλει να δούμε πάλι τα σύνορα του παρελθόντος που πρέπει να προσθέσω ότι ίσχυαν κυρίως για λόγους ασφαλείας. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει προοδεύσει πάρα πολύ και αν επισκεφτείτε την περιοχή θα δείτε πόσο έχουμε προχωρήσει. Δεν θέλουμε να οπισθοδρομήσουμε. Άκουσα την παρουσίαση του Δ. Φίνεμορ και της ε, Δ. Χέιουαρτ. Μιλήσατε για πιθανότατα διαφορετικούς κανόνες για τη Βόρεια Ιρλανδία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους κανόνες για την συνεργασία δύο κυρίαρχων μελών και σε κανόνες ε, που θα πάψουν να ισχύουν ε, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις διαφορές. Με ενδιαφέρει η μελέτη σας, διότι δεν κοιτάτε συγκεκριμένα τις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και το υπόλοιπο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Δόκτωρ Χέιγορντ, ε, Κυριακή βράδυ, ε, έβαλε κάποια στοιχεία στο Twitter, τα οποία ήταν πολύ χρήσιμα. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να τα κοιτάξουμε. Τα στοιχεία αυτά μας λένε ότι το 60% των εξωτερικών πωλήσεων ε, της Βόρειας Ιρλανδίας ε, έχουν ε, προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, το 60%. Το 15% του εμπορίου πραγματοποιείται με την Ιρλανδία το 16% με το υπόλοιπο του κόσμου και 9% με το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε λοιπόν ότι η σημαντικότερη αγορά για μας είναι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Το να ε, ε κλείσετε σε μια ξεχωριστή ε, ζώνη εμπορίου, να μας απομονώσετε από την πιο σημαντική αγορά για μας, ε, δεν είναι μόνο πολιτικά απαράδεκτο, θα αποτελέσει καταστροφή οικονομική. Έχω και πολλές άλλες παρατηρήσεις, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα συναντηθώ με τον δόκτωρα Φένιμορ για να το συζητήσουμε ε, ε, ότι θα έχουμε άλλες ευκαιρίες. Και στον ε, κύριο Λάγκ θα ήθελα να πω ότι με εκπλήσει η μεροληπτική στάση στην εκθεσή σας. Όταν διαβάζω ότι όσοι ψήφισαν να αποχωρήσουν ε, ε, από, την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βασίζονταν σε προκαταλήψεις και νοσταλγικές ιδέες. Τι να σας πω, πρόκειται για δημοκρατική απόφαση των ψηφοφόρων του Ηνωμένου Βασιλείου και νομίζω ότι είναι απαράδεκτος ο τρόπος που το περιγράφεται. Πάλι αναφέρεστε στο κόμμα μας, ε, το Δημοκρατικό Κόμμα των ε, Ενωτικών, αναφέρεστε στη συμφωνία του Μπέλφαστ και λέτε Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρόσφατη δικαστική υπόθεση στη Βόρεια Ιρλανδία. Και μάλιστα κάποια επιχειρήματα δεν ε, ακούστηκαν όσον αφορά την ε, ασφάλεια τροφοδοσίας, ε, διότι θεώρησαν ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη συμφωνία του Belfast. Στο συνάδελφο που μας υποβάλλει κάποιες λύσεις για τα τελωνιακά ζητήματα, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί επικοδομητικές και καινοτόμε λύσεις. Ε, αυτή εδώ πέρα, αυτό είναι ένα πρώτο παράδειγμα μιας τέτοια ευέλικτη και καινοτόμας λύσης. Πρόεδρο. Ε, πρέπει να κλείσω το κατάλογο των, των μιλητών. Ε, δύο λεπτά αναομιλητή, δέκα ομιλητέ έχουμε. Σα παρακαλώ λοιπόν επικεντρωθείτε στι ερωτήσει που θέλετε να θέσετε και να είσαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Με δύο λεπτά θα δώσουμε το λόγο σε όλους και θα μπορέσουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Η Μαρτίνα Άντερσον. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σήμερα εδώ για την παρουσία σας. Και τι λυπάμαι που έχασα το ξεκίνημα της, την αρχή της παρουσίασής σου από το Λονδίνο. Έρχομαι όπου ξεκινήσαμε ε, την ε, εκδήλωση για να δείξουμε πώς ε, είναι δυνατόν να έχουμε ειδικό καθεστώς για την Βόρεια Ιρλανδία εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Ντέιβιτ σχετικά με την διαφοροποιημένη προσέγγιση και την εδαφική διαφοροποίηση, διότι Αυτό είναι κάτι που έχει αναφερθεί. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές ε, όπως για την ε, Γρυλανδία. Ενδιαφέρον ε, είναι στην έκθεσή σας ότι θεωρείτε ότι η σταθεροποίηση απορρέει από τη συμφωνία του της Μεγάλης Παρασκευής, αναφέρεστε στα δικαιώματα, δεν θέλουμε ε, επιδείνωση όσον αφορά τα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν είναι ευρύτερη η προσέγγισή σας. Η Επιτροπή μας ε, νομίζω ότι έχει καταλάβει πια τι σημαίνει, πόσο σημαντική είναι η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Όσον αφορά τα εφή σύνορα, θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο, εάν δεν πρόκειτο για μια χώρα ε, διχασμένη που βγαίνει επιτέλους από μια σύγκρουση. Όλα ωραία και καλά, αλλά η πρότασή σας ε, για τα ευφυή e e σύνορα είναι ε, ανόητη η συνοριακή πρόταση ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να λειτουργούσε αυτό σε άλλη περίπτωση, αλλά δεν θα λειτουργήσει στην Ιρλανδία. Επίσης, Τζον αναφέρθηκε στο τι σκοπεύει να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, όσον αφορά το, την γεωργία, αλλά πολλοί αγρότες στον Βορρά θα θεωρήσουν ότι αυτό θα είναι επιζήμιο για αυτούς. Α είμαστε σαφείς. Ε, μίλησε για επιδείνωση των μέτρων για την υγεία των ζώων. Εάν όμως ε, δεν είχαμε τέτοια μέτρα, δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα του καταρροϊκού πυρετού των εγωπροβάτων. το 60% των ε, ε, ενωτικών ε, εξετάζουν το θέμα των συνόρων και 562 προβουλευτέ εδώ στο Κοινοβούλιο θεώρησαν ότι η Βορεια Ιρλανδία θα πρέπει να παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά Αυτός ε, θα είναι ο, μόνο τρόπο, ο μόνος τρόπος να έχουμε τα ε, ρυθμιστικά πρότυπα και να μην έχουμε επιστοχώρηση σε σχέση με την ε, Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Ως Κοινοβούλιο, λοιπόν, θα πρέπει να επιμείνουμε στην συνέχιση της ισχύω της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής όσον αφορά όλες τις πτυχές της. Και το θέμα δεν είναι μόνο τα σύνορα, είναι η σταθερότητα, είναι τα δικαιώματα η μη επιδείνωση των δικαιωμάτων και νομίζω ότι η Επιτροπή μας ε, έχει ε, πιάσει όλες τις Σε Συγγνώμη που ε, ξεπέρασα το χρόνο μου, αλλά καταλαβαίνετε ότι το θέμα αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Επιμένω στα δύο λεπτά. Η Μερσέντες Μπρέσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Προφανώς και η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις σας, αλλά το θέμα είναι ε, ότι να κατανοήσουμε ποιες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο εύκολα σημαίνει να ε, γνωρίζουμε και τι προτείνει επισήμως το Ηνωμένο Βασίλειο για την κατάσταση στην Ιρλανδία. Μια πρώτη ερώτηση στον καθηγητή Λάρσον για τα έξυπνα σύνορα. Το πρόβλημα είναι ότι μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας Προφανώς και υπάρχει ευρωπαϊκό σύνορο, αλλά η Νορβηγία συμμετέχει και στον ε, ε, Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στον ΕΟΧ και νομίζω ότι είναι και τμήμα της Σέγγεν. Επομένως είναι πολύ πιο εύκολη η διαχείριση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι και εύκολη η διαχείριση ε, στην περίπτωση κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν δεν δεχτεί καμία διάκριση και συμπεριλάβει και τη Βόρεια Ιρλανδία στην έξοδο από την ε, Τελωνιακή Ένωση και από την είναι αγορά, διότι σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη ε, και δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε τόσο εύκολα. Όσον αφορά τους υπολείπους, ε, η ερώτηση αντιστρέφεται. Πώς θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να εγγυηθούμε τις ε, συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής χωρίς σύνορα, εκτός και αν παραμείνει όλο το ε, Ηνωμένο Βασίλειο εντός της τελωνιακής ενίωσης και της ενιαίας αγοράς, ίσως ε, με κάποιες ε, διαφορές και έχουμε περισσότερο ελβετικό μοντέλο και όχι μοντέλο ΕΟΧ. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τίθεται θέμα συνόρου. Εάν δεν γίνει αυτό, πώς φαντάζεστε μια κατάσταση στην οποία γίνονται σεβαστοί οι πυλώνες της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εγγυηθούμε και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευράς ε, ε διέλευσης εμπορευμάτων, διότι αν υπάρχει σύνορο εκεί, ε, το οποίο ε, σημαίνει ότι θα είναι και τελωνιακό σύνορα με κάθε σημασία ε, του όρου σημαίνει ότι πρέπει κάπως να διαχειριστούμε αυτά τα σύνορα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορούμε να βρούμε μια έξυπνη λύση για να αντιμετωπίσουμε ε, την περίπτωση μιας πλήρης εξόδου της Τελωνιακής Ένωσης από την Τελωνιακή Ένωση και την ενή αγορά, δηλαδή δεν θα υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ε, ανθρώπων, εμπορευμάτων και κεφαλαίου, δηλαδή των τεσσάρων ελευθεριών. Ευχαριστώ. Ashley Φόξ, αλλά θα ήθελα να σας ε, προειδοποιήσω, θα χρησιμοποιήσω το σφυράκι μου μετά από τα δύο λεπτά. Εντάξει, θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένο, κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω τους δόκτωρες Hayward και Φίνεμον για την παρουσίαση. Όπως ξέρετε, η Βρετανική κυβέρνηση δεσμεύεται στην τήρηση τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και θέλει να ε, ε, διαπραγματευτεί μια βαθιά και ειδική εταιρική σχέση με τους νέους γείτονες. Εσείς αναφέρεστε στην ε, ίση ισχύ των δύο παραδόσεων στη Βόρεια Ιρλανδία. Ακούσαμε δύο φωνές σήμερα το απόγευμα και λέτε ότι θα πρέπει να την χάνουν αντίστοιχου σεβασμού επειδή και οι δύο πλευρές θέλουν να εξασφαλίσουν ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη η λειτουργία των συνόρων και θα είναι προσπελάσματα τα σύνορα. Όταν αναφέρεστε σε προτιμησιακή μεταχείριση, δεν βγαίνει κανένα νόημα ούτε από οικονομική σκοπιά, όπω είπατε, αλλά προσβάλλει και μία από τι δύο αυτέ παραδόσει και παραβιάζει τη συνταγματική ακαιρεότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να με εξηγήσετε γιατί θεωρείτε ότι η προσβολή μια παράδοση είναι αποδεκτό στην προτινόμενη λύση σα, αλλά όχι της άλλη. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα επ' αυτού. Κύριε Κάρστον, ε, σας ευχαριστώ για την εκθεσή σας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Χρειαζόμαστε μια έξυπνη, ομαλή και ασφαλή οδό για να έχουμε ε, ε, αόρατα σύνορα όπως ελπίζουμε. Δεν είπατε τίποτα όσον αφορά το χρονοδιαγράμματα, αλλά έστω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2019 και θα υπάρχει μια διετής μεταβατική περίοδο. Έχετε λοιπόν το Μάρτιο του 2021 συγγνώμη, ως καταληκτική ημερομηνία. Πότε πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή αυτών των έξυπνων συνόρων. Και ένα σχόλιο για τον ε, κύριο Λάγκ. και εγώ απογοητεύτηκα από την παρατηρησία σας όταν είπατε και παραθέτω ότι η απόφαση αποχώρηση δεν ήταν αποτέλεσμα μια ε, προσεκτική αξιολόγηση από τι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μια διολογική επιλογή που βασίζεται σε προκατάληψη, άγνοια και νοσταλγία. Επειδή εγώ είμαι εξ αυτών που έκαναν εκστρατεία για παραμονή, νομίζω ότι η δική σα η άγνοια και η προκατάληψη είναι αυτέ οι οποίε προβάλλονται και είναι λυπηρό να ακούγουμε τέτοιε παρεμβάσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλεια, που και θέσετε και την ερώτησή μου. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω, κύριε Κάλσον, ότι αυτό ο χρονικό παράγοντα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, Συμπρόεδρε, και πρέπει να σας πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ οι παρουσιάσεις που έγιναν σήμερα. Ήθελα να σας πω ότι στα όσα είπαν οι εκπρόσωποι του Queen's University στο Belfast, έχω την εντύπωση πως η δική σας λύση έχει να κάνει με κανονιστική ισοδυναμία και Για τα όσα προκύπτουν από, τη δεύτερη, το δεύτερο σκέλος της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής για τα, το κανονιστικό πλαίσιο, θα ήθελα να πείτε το εξή, Πιστεύετε εσείς πως όπου λειτουργούμε στα πλαίσια της βάσης και του άξονα και στα πλαίσια της συμφωνίας, με τους φορείς που βρίσκονται και από τις δύο πλευρές των συνόρων, θα μπορούσαμε εκεί να ενισχύσουμε ή να, ε, να, να ισχύσουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υπάρχουν τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη στιγμή που μεταγράφουν μεγάλα κομμάτια του κανονισμού που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στη Σκωτία για παράδειγμα, που εφαρμόζεται στη Σκωτία και δεν εφαρμόζονται κάπου αλλού. Που αυτή τη στιγμή αν είχαμε μια κυβέρνηση στην αποκεντρωμένη βουλή της Βορείου Ιρλανδίας θα μπορούσε να γίνει εκεί η μεταγραφή που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβέρνηση από τη στιγμή που έχει εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα κάποιο από τι Βρυξέλλε. Δηλαδή, σε αυτού του ορισμένου χώρου, στα πλαίσια τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να έχουμε κανονισμού ευρωπαϊκού ε, που να ισχύουν και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία είναι αναλυτικά δυτικά. Ανατολή Δύση, που είναι το μεγάλο κομμάτι τη εμπορία από την ε, Ιρλανδία, να ισχύουν οι κανονισμοί της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή, έτσι ώστε η Βόρεια Ιρλανδία να έχει ε, τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ε, και τις δυνατότητες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις νέες δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πρέπει να σας πω ότι για την εγκληματικότητα και τα λοιπά συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τέμπλ Λαν. Ξέρουμε, ξέρουμε, θυμόμαστε το παρελθόν. Όπου υπάρχουν σκληρά σύνορα, έχουμε λαθρεμπόριο, έχουμε παραστρατιωτικές ομάδες, το ξέρουμε αυτό, το ξέρει ε, και η κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία ε, στην ε, Δημοκρατία της Ιρλανδίας και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο για το μέλλον γιατί γνωρίζουμε δυστυχώς ποια ήταν η κατάσταση στο παρελθόν. Ο Μπράιν Σαντλή to the speakers. Ο Σον Κέλλη, με συγχωρείτε. Ακούσαμε πολλά και είναι δημιουργικές και ευφυείς λύσεις με πολύ λίγες λεπτομέρειες προσπάθησατε να μας προσφέρετε κάποιες λύσεις. Και, εν πάση μπορούν να αποτελέσουν μια αφετηρία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τα ευφυή e σύνορα. Και τη δυνατότητα ε, να πετύχουμε το ιδανικό που είναι ότι τα σύνορα ενώνουν, συγγνώμη, τα σύνορα χωρίζουν, τα τελωνία ενώνουν γιατί νομίζω ότι πρόκειται να εισαχθούν σύνορα μεταξύ Δημοκρατίας Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας, οπότε κάποιο είδους ε, τελωνιακά ζητήματα θα προκύπτουν. Τα παραδείγματα που δώσατε δεν νομίζω ότι είναι απολύτω κατάλληλα, αλλά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία είναι δύο ξεχωριστέ χώρε. Καναδά, Ηνωμένε Πολιτείε, δύο διαφορετικέ χώρε. Σουηδία, Νορβηγία, ίσως εφαρμόζεται καλύτερα στη δική μας περίπτωση, αλλά δεδομένου πως το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να εγκαταλείψει και την ενιαία αγορά και την τελωνιακή ένωση, δεν είμαι σίγουρος πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι τέτοιο, αλλά θα ήθελα να μας πείτε τι θα μπορούσε να λειτουργήσει στα πλαίσια των ευφυών συνόρων. ελευθερία κυκλοφορίας ατόμων, αγαθών. Και τι δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε εάν το χειρότερο σενάριο ε, εφαρμοστεί και φύγει και από την Τελωνιακή Ένωση και την Ενιαία Αγορά του Ενωμένου Βασίλειου. Και σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που προσπαθείτε να δώσετε λεπτομέρειες για, τους, ε, για το πλαίσιο που όλοι περιγράφουν χωρίς λεπτομέρειες το τελευταίο ε, διάστημα. Ο κύριος Σίλβα Περέιρα, τελευταίος ομιλητής. Μία ερώτηση μόνο. Κύριε Κάρσεν, ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων. Μόνο γι' αυτό. Καταρχήν συγχαρητήρια για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και έξυπνη έκθεση. Αλλά χρειάζομαι μια διευκρίνηση. Δεν προτείνεται αόρατα σύνορα προτείνεται φυσικά σύνορα που θα ελέγχεται, που θα ελέγχονται. Γιατί αν κατάλαβα καλά, η πρότασή σας είναι να έχουμε ελευθερία κυκλοφορίας ατόμων που καλύπτονται από το κοινό χώρο ε, διελεύσεων και οι υπόλοιποι θα χρειάζεται να πηγαίνουν στα σύνορα, στα συγκεκριμένα σημεία και εκεί θα απαιτείται να δείξουν διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο Οπότε είναι ένα χαλαρό σύνορο στα πλαίσια του δυνατού. Δηλαδή θα έχουμε και σύνορα και συνοριακούς ελέγχους για όσους δεν ε, καλύπτονται από το Common Travel Area. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακίνες. Ο κύριος Μακίνες. κυρία Μακίνες. Ας μπω στο ψητό, αγαπητοί συνάδελφοι. Το βασικό είναι το πλαίσιο. Στις δύο παρουσιάσεις, εντάξει, το είχαμε. Στην τρίτη είχαμε απλώς λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, ευφυείς σύνορα, ευφυείς λαθρέμποροι. Έχουμε μακρά και λυπηρή παράδοση πολύ έξυπνων λαθρεμπόρων στην περιοχή μας. Σας τα αποφύγουμε λοιπόν αυτά, αλλά για να μιλήσω λίγο πιο σοβαρά. Εγώ στάθηκα ακριβώς πάνω στα σύνορα και από τις δύο πλευρές, με το κρύο, με πραγματικό κόσμο, ε, ε, την περασμένη εβδομάδα και ο κόσμος αυτός φοβάται. Ένας μου είπε ότι εγώ ήθελα να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τι θα γίνει τώρα. Και άλλος είπε, στη δική μου ε, εκλογική περιφέρεια, εμεί ξέρουμε ε, ποια θα είναι τα αποτελέσματα και δεν ήθελα. Και ξέρουμε τι είπαν και στην Επιτροπή ΕΜΒΗ. Γιατί υπάρχουν περιβαλλοντικά θέματα, θέματα ασφάλειας τροφίμων και όλα αυτά ε, προκύπτουν λόγω Brexit. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε τις πολιτικές συνέπειες του Brexit και παρόλο που σέβομαι αυτούς οι οποίοι παρουσιάζουν τεχνικές λύσεις, τεχνικές λύσεις δεν επαρκούν όταν το πρόβλημα είναι πολιτικό. Έχουμε ένα κομμάτι του νησιού της Ιρλανδίας που είναι κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά εμείς στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας είμαστε τμήμα της ειρηνευτικής διαδικασίας. Και έχω τη συνάδελφο με την οποία συνεργάζομαι ε, στην Επιτροπή και θα έλεγα στην Ταϊάν που είναι από το DUP πως ναι, είσαι υπεύθυνη πολιτικός και έχεις μια ιδιαίτερη ευθύνη αυτή τη στιγμή ως μέλος του DUP να χρησιμοποιήσεις την επιρροή που έχεις, που είναι τεράστια στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και να τους πεις βρείτε μια λύση η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τις πολιτικές ευαισθησίες από όλες τις πλευρές. Γιατί και οι δικοί σας Γεωργοί είναι σαν τους δικούς μας. Θέλουν βεβαιότητα, ασφάλεια, δεν θέλουν διαταραχή, φόβο, αβεβαιότητα. Και αυτό κυριαρχεί επί τόπου σήμερα. Και αυτό που έκανε ήταν δήλωση, συνάδελφοι, δεν ήταν ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, οι λαθρέμποροι πολύ συχνά βρίσκονται μπροστά από ε, το σύστημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε δεν είναι βέβαιο ότι όλες οι αρμοδιότητες θα επιστρέψουν αυτομάτως ε, στα διάφορα κοινοβούλια. Επίσης, ε, δεν... Επίσης, μπορούμε να συγκρίνουμε με τα σύνορα Νορβηγίας-Σουηδίας, ε, διότι η Νορβηγία είναι μέλος της του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων ε, είναι και αυτό ένα θέμα. Όσον αφορά το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα, ε, το, τα του 2015 προειδοποίησα για το θέμα αυτό, ε, αλλά το DUP ισχυρίστηκε ότι αυτό θα είναι διμερές θέμα ανάμεσα στο Λονδίνο και το Δουβλίνο και ότι δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, υπάρχει ένα μέρος του Βρετανικού εδάφους ε, που θα παραμείνει στην Τελωνιακή ε, Ένωση μετά το Brexit ε, και αναφέρομαι στην Κύπρο, τις βάσεις στην Κύπρο που θα παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την συνθήκη θα συμμετέχουν και στην ενιαία αγορά. Εγώ πάντως υποστηρίζω ότι αυτή η συνθήκη ε, συνεπάγεται και η ηθική υποχρέωση να ε, έχουμε σωστή διαχείριση των συνόρων στην Ιρλανδία. Και θα πρέπει να λύσουμε το θέμα αυτό με δημοκρατικό τρόπο, πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή το DUP έχει τη θέση που έχει και που έχουμε κυβέρνηση μειονότητα ε, στην Ιρλανδία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, δημοψήφισμα στην ε, Βόρεια Ιρλανδία και να δούμε, διότι εάν πιστεύουμε στην δημοκρατία θα πρέπει να έχουμε μια κυρίαρχη απόφαση εκεί. Πρόεδρος, ε, δεν νομίζω ότι, έχει, ότι υπάρχει πολύ εμπορική δραστηριότητα στις στρατιωτικές βάσει τη Κύπρου, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι για τα συνορα σουηδια Σουηδίας-Νορβηγίας ε, που είναι ό,τι εγκύτερο έχουμε σε ξυπνά σύνορα ε, με συγκρίσιμους όρους. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ακόμα και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία διέλευση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, οχήματα με ε, φυσικούς ελέγχους. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε κατά πόσο ισχύει. Ορισμένες φορές υπάρχουν και πολύ σημαντικέ καθυστερήσει. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξή. Πολλέ από τι συζητήσει μα ε, βασίζονται στην υπόθεση ότι ε, κατ' ουσίαν ε, θα διαπραγματευτούμε και μία συμφωνία, διότι οποιαδήποτε λύση θα είναι αποτελεσματική μόνο αν συνεργαστούν όλοι και γίνει από κοινού. Η ερώτησή μου είναι τι γίνεται σε περίπτωση που έχουμε εκδοχές τις οποίες δεν υπάρχει συνεργασία. Μια τριώτη περίπτωση, ειναι τι γινεται σε περιπτωση που εχουμε εκδοχες τι οποιες δεν υπαρχει συνεργασια μια περιπτωση πρωτη περιπτωση να μην υπάρξει συμφωνία για ε, το διαζύγιο, μια κατάλληλη συμφωνία διαζυγίου, γιατί να μην λησμονούμε ότι κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση έχουν εξετάσει και αυτό το ενδεχόμενο και θα φαντάζεται κανείς ότι κάποιοι θέλουν και να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι έστω ότι όλα είναι σωστά, υπάρχει συμφωνία, αλλά πέντε χρόνια αργότερα υπάρχει μια φυτογενομική κρίση. Ή για παράδειγμα θυμηθείτε τις τρελές αγελάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της φύσεως αυτού. Θυμάστε τι συνέβη πριν από 20 χρόνια. Υπήρχε κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, παρά το γεγονό ότι ήταν τότε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ε, υπό Τζον Μέιτζορ ε, είχε μια πολιτική μη συνεργασία με την Ευρώπη και γι' αυτό αλλά και για ένα θέματα. Ε, υπήρχε η ε, ε, το αρκτικό λέξο PONHCE, PONS, ε, ε, και θα έπρεπε να ληφθούν ισχυρά στατευτικά μέτρα εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσουν ε, τις τρελές αγελάδες ή οτιδήποτε άλλο να μην περάσουν και θα χρειαστεί συνδρομή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει κάποια άλλη λύση που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Τελευταίος ο μιλητής η Τζάιάν Τζέιμς και μετά θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η πεποίθησή μου είναι ότι τα Ιρλανδικά θέματα είναι θέμα που αφορά το Δουβλίνο και το Λονδίνο και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσά δεν αρέσκεστε να τα ακούτε αυτό. Μου άρεσε η έκθεση για τα σύνορα, ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη, πολύ ενημερωτική και είχε πολύ σημαντικά στοιχεία. Και ίσως ε, αυτό που πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν και είναι και η αίσθηση της ερώτησής μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σε τεχνολογίες έξυπνων σύνορων στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και σε άλλους τομείς ε, σε άλλε περιοχές όπου υπήρχαν προβλήματα με μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες, πρόσφυγες, ε, ετούντες άσυλο, αυθεντικού σημείου. Γιατί λοιπόν αυτή η τεχνολογία και η εφαρμογή τη που θα μπορούσε να ε, είναι λύση του προβλήματος αγνοείται στη μία περιοχή και προωθείται σε μια άλλη περιοχή. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω ε, ότι η Πρωθυπουργό μα, το Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, η κυρία Τερέζα Μέη, είπε ότι δεν θα υπάρχουν σκληρά σύνορα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οποιοδήποτε σκληρά σύνορα θα τα υψώσει η Ιρλανδική πλευρά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω ποιο από εσά θέλει να απαντήσει. Εσεί ε, θα αποφασίσετε ποιο θα μιλήσετε πρώτο και με ποια σειρά σα. Δίνω το λόγο να επιλέξετε. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που κάνατε και θα μιλήσω στο το δυνατόν πιο σύντομα. Θα ξεκινήσω τις ερωτήσεις από τα όσα είπε η Νταϊάν Τότς, μετά ο κύριος Φόξ. Και θα συνεχίσω με τους υπόλοιπους. Οι προτάσεις μας βασίζονται στην αρχή πως η Βόρεια Ιρλανδία θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και πως το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι κυρίαρχο και δεν θα υπάρχει καμία διάκριση ή προκατάληψη εναντίον των διαφορετικών πολιτικών προσδικιών που έχουν ε, οι άνθρωποι στη Βόρεια Ιρλανδία. Η διαφοροποίηση δεν έχει να κάνει με τη συνταγματική ε, ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό είναι πολύ βασικό στο να διατηρηθεί συμφωνία. Δηλαδή, όπου δεν είδε θίγεται αυτή η αρχή. Αυτή η διαφοροποίηση υπάρχει ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αν η Βόρειος Ιρλανδία έχει διαφοροποιημένες διευθετήσεις έτσι ώστε να συνεχιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία στο νησί της Ιρλανδίας, αυτό δεν υποσκάπτει τη συνταγματική ακαιρεότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να προτείνουμε τρόπους, όπως είπαμε πολύ ανοιχτά, η Βόρεια Ιρλανδία να έχει το καλύτερο και από τις δύο περιπτώσεις ευελιξία, φαντασία. Και αυτή είναι μια μοναδική περίπτωση να στηρίξουμε και ευκαιρία να στηρίξουμε τη συμφωνία. Οπότε η επιλογή δεν είναι ή πιο κοντά ε, στη Βρετανία ή πιο κοντά στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Χρειάζεται μια λύση με ευελιξία, με φαντασία, με διαφθετήσεις τις οποίες θα ισχύσουν στη Βόρεια Ιρλανδία έτσι ώστε να έχει το καλύτερο από όλα τα σενάρια. Και είναι αξιοσημείωτο πως το μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορίου στην ε, Βόρειο Ιρλανδία είναι εσωτερική, εσωτερικό εμπόριο. Είναι μια οικονομία όχι πολύ αναπτυγμένη και οι περισσότερες πωλήσει φεύγουν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, και πάλι εδώ δεν πρέπει να χρειαστεί να επιλέξουμε μεταξύ αυτών των πωλήσεων και πωλήσεων στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρκετά αξιοσημείωτο πως η επιλογή είναι τώρα το να επιστρέψουμε σε ε, σε μια κατάσταση όπου όλες μας οι αγορές και το εμπόριο θα πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και να χάσουμε αυτό το 24-25% που πηγαίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πρέπει να βρούμε κάποια ε, ευέλικτη λύση και, φαντα... και φάνταστη λύση για να καταφέρουμε ακριβώς αυτή η διαφοροποίηση να εξασφαλιστεί. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σας, η κυρία Hayward. Θέλω να τονίσω πως αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε η Βόρεια Ιρλανδία να στραφεί σε μια εναλλακτική αγορά. Όχι. Θέλουμε να βρούμε μια λύση που θα τη επιτρέψει να διατηρήσει την βαθιά ε, ολοκλήρωση την οικονομική με το Ηνωμένο Βασίλειο και παράλληλα να τη διευκολύνει να διατηρήσει το δυνατόν περισσότερο το status quo στο νησί τη Ιρλανδία. Και αυτό σημαίνει συνέχιση ε, ουσιαστικά τη συμφωνία τη μεγάλη παρασκευή και θα συμφωνήσω με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι εδώ. Υπάρχει ευελιξία στο Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου ε, υπάρχουν οι δυνατότητες της αποκεντρωμένης διοίκησης και νομίζω ότι στο Σύνταγμα μέσα προβλέπονται τρόποι έτσι ώστε η διαταρχή που θα δημιουργήσει αναμφίβολα το Brexit στο νησί της Ιρλανδίας να μείνει σε ένα ελάχιστο δυνατό. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ε, καταρχάς να υπογραμμίσω κάτι που γράφω στην έκθεση και που είπα και στην παρουσίασή μου. Τα τρία παραδείγματα που χρησιμοποίησα στην έκθεση δεν είναι τέλεια παραδείγματα, ε, αλλά το θέμα εδώ είναι ότι κάθε ε, λύση μπορεί περιέχει στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια πιο ευφυή επιλογή. Και όσον αφορά την ε, τελευταία ερώτηση ε, για την, ε, τα σύνορα Νορβηγίας-Σουηδίας, φυσικά υπάρχουν διαφορές, αλλά υπάρχουν και εκεί κάποια πράγματα που δεν έχουν εφαρμοστεί, τα οποία μπορούν όμως να εφαρμοστούν εδώ πέρα. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν να σχετικοποιήσουμε το γεγονός ότι η Νορβηγία, η Σουηδία δεν είναι το τέλειο παράδειγμα. Ε, η Σουηδία, Νορβηγία είναι, ας το πούμε έτσι, η λύση 1.5, ε, ενώ εμείς ε, φτάνουμε στο 2.0 στην Βόρεια Ιρλανδία. Λέω απλά δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στη λύση αυτή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εδώ πέρα και πολλά εξαρτώνται από ε, το πώς λειτουργούν τα τελωνία και μάλιστα τα στοιχεία αυτά συνήθως ε, δεν είναι ορατά. Διευκολύνουν το εμπόριο, στηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και πολλά από τα θέματα αυτά μοιάζουν με την περίπτωση την οποία συζητάμε εδώ. Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες, υπάρχουν στοιχεία, θα πρέπει όμως ε, να βρούμε μία σύγχρονη επιλογή. Ο παράγοντας του χρόνου φυσικά είναι πολύ σημαντικός ε, και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα, σήμερα. Ίσως θε ολότελα, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν. Ίσως λοιπόν να ξεκινήσουμε αύριο. Ε, να κάνω μια εκτίμηση όμως, η επαγγελματική μου θέση είναι ότι εντός της διετίας θα είναι δυνατόν να έχουμε μια ρύθμιση. Δεν θα είναι τέλεια, θα είναι μια πρώτη εκδοχή Μπορεί όμως να υπάρξει και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία αναφέρω υπάρχουν ήδη στην Ιρλανδία, Βορεια Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκοπός είναι να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν, να τα αναβαθμίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία ώστε να λειτουργούν καλύτερα από ό,τι σήμερα. Ώστε να έχουμε σύνορα τριβέ. Ε, η κοινή περιοχή, το CTA, το Common Travel Area, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όμως σε συνδυασμό με προγράμματα ε, ταξιδιωτών εμπιστοσύνης, κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και ε, εάν ε, δεν εμπίπτει κανείς ένα τέτοιο πρόγραμμα, ίσως να πρέπει να περάσει σε συγκεκριμένο σημείο διέλευσης των συνόρων. Θέλουμε να αποφύγουμε τις ουρές και από τις δύο πλευρές των συνόρων, τη συμφόρηση και για τους, και για τους ε, ανθρώπους ε, και για τα αγαθά. Όσον αφορά το θέμα των ε, λαθρεμπόρων, επί πολλά χρόνια προσπαθώ να καταπολεμήσω το έγκλημα και τους λαθρεμπόρους που ήδη δραστηριοποιούνται και σε άλλα μέρη της Ιλλανδίας. Κάνουν τη δουλειά τους ήδη τώρα. Ο καλύτερος τρόπος που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα με τις διάφορες μορφές που παίρνει, όπως γίνεται για παράδειγμα αυτή την στιγμή στα σύνορα της Βραζιλίας. Ε, το κυριότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Θα υπάρχει ανάγκη λοιπόν για αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και από διάφορους ε, οργανισμούς. Ε, εάν λοιπόν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό χωρίς να καθυστερήσουμε τις μετακινήσεις ε, ανθρώπων και αγαθών, ε, αυτό θα είναι καλό. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις πληροφορίες που έχουμε και τις μυστικές πληροφορίες για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Πιστέψτε με, τα προβλήματα αυτά ήδη υπάρχουν. Αυτή τουλάχιστον είναι η επαγγελματική μου θέση. Νομίζω ότι αυτά τα διαφορετικά στοιχεία μπορούμε να τα συνδυάσουμε, να ε, καταφέρουμε να έχουμε ένα σύστημα που θα λειτουργήσει ε, και μάλιστα εντό του χρονοδιαγράμματο. Αλλά βέβαια δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και γι' αυτό μία από τι τελευταίε μου παρατηρήσει εδώ πέρα είναι ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε το γεγονό ότι άσχετα από το τι μορφή θα έχει το σύνορο θα πρέπει να υπάρξει διαχείριση του σύνορου. και αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο ουδέτερο ως προς το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε, και περίπτωση σκληρού Brexit και σε ε, περίπτωση ενός πιο ήπιου Brexit και θα πρέπει να ε, υπάρχει σε δύο χρόνια και ε, επίσης θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως ε, να μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα και να διευκολύνει το εμπόριο. Η λύση που έχουμε εδώ πέρα νομίζω ότι ε, Υπάρχουν εδώ κάποιες ειδικέ περιστάσεις, το αναγνωρίζω αυτό. Κάποιοι αναφέρθηκαν στην πολιτική κατάσταση, εγώ ε, προτίμησα να μην το κάνω. Νομίζω όμως ότι μια τεχνική λύση μπορεί να μας βοηθήσει και στην εξέβρεση πολιτικής λύσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, υποθέτουμε ότι το πρόβλημα στα σύνορα σχετίζεται με τα τελωνία. Πολλοί από τους ε, ελέγχους ε, όμως θα σχετίζονται με την ε, εσωτερική αγορά, όπως για παράδειγμα η ασφάλεια των τροφίμων. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο οι δασμοί, αυτό μάλλον είναι μια από τις πιο εύκολες πτυχές. Δεν ξέρω αν ασχολείστε και με αυτό. Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς ε, χρειάζεται να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο βασίζεται στην γνώση των ε, εμπόρων. Ακόμα και όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα προγράμματα ε, έμπιστων εμπόρων και ταξιδιωτών εμπιστοσύνης θα πρέπει να εφαρμοστούν άσχετα από το τι τελικά προταθεί και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ε, ότι ε, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον ε, ενωσιακό τελωνιακό κώδικα. Θα είναι νομίζω δυνατόν να βρούμε μια λύση που να ευθυγραμμίζεται με τον ενωσιακό τελωνιακό κώδικα και τα διεθνή πρότυπα. και τα δύο μέρη εδώ θα πρέπει να διαπραγματευτούν ε, εμπορικές συμφωνίες ε, με άλλα μέρη του κόσμου. Με τη συγκεκριμένη λύση λοιπόν θα είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο ε, οι δασμοί και οι φόροι, υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν. Ευχαριστώ, καθηγητή Στέμπριλα. Ένα σχόλιο μόνο οποιοδήποτε πιστεύει ότι η ιδέα που προτείνεται ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να έχει δικό της χώρο ελευθέρων εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκοπεί η οικονομία της Βόρειας Ιρλανδίας από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ακριβής περιγραφή των συνεπειών και σε καμία περίπτωση